Hello everyone. If you take your seats, then we can uh, start our meeting today. Καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρώτα θα δώσουμε το μικρόφωνο στους διερμηνείς, διότι θέλουν να κάνουν μια ανακοίνωση. Παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας και βάλτε το αντίστοιχο κανάλι της γλώσσας σας.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 Η COP24, διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, στην Κατεβίτσε, στην Πολωνία, από 3 έως 12 Δεκεμβρίου. Έχουμε λάβει τους συνεισηγητές και θα τους δώσω το λόγο. Okay, so first I'll make Πρώτα θα κάνω εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Από την υπογραφή της Συμφωνίας των Παρισίων και την κύρωσή της ε, και μάλιστα σε ένα ρυθμό χωρίς προηγούμενο. Η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η εφαρμογή των ε, εθνικών δεσμεύσεων και να συνεχίσουμε φυσικά να προχωρούμε. Έχουμε δείξει τη δέσμευσή μας τους ε, τελευταίους μήνες με τη Συμφωνία για τη Δέσμη Μέτρων για το Κλίμα και πιο πρόσφατα στα όσα έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Καθαρή Ενέργεια. Παρά τις θετικές εξελίξεις ε, και παρά το γεγονός ότι η ρυθμοί αυτοί δεν εγγυώνται ότι θα έχουμε σημαντική ε, αντιστροφή του κλίματος. Ε, γι' αυτό ακριβώς χαιρόμαστε που θα ε, έχουμε το φθινόπορο τον οδικό χάρτη μέχρι το 2050 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αναβάθμιση των στόχων μέχρι το 2020 μετά από το διάλογο ο οποίος θα γίνει πέραν των εσωτερικών μας δράσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε όλους τους τομείς να συμβάλλουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια, ιδιαίτερα το τομέα της ε, ναυτιλίας και της αεροπορίας, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα σε εξωτερικό επίπεδο. Μπορούμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην χρηματοδότηση του κλίματος ε, και επίσης ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην διεθνή κλιματική διπλωματία. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των ε, μη κρατικών ε, παραγόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτά όλα φυσικά είναι βασικά στοιχεία τα οποία έχουμε τονίσει σε αυτό το κοινό ε, ψήφισμα. Είμαι βέβαιη ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν πολλά να προσθέσουν και αυτό και θα κάνουμε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν και στις διαπραγματεύσεις στην Κατοβίτσε. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδόλφους και πρώτα-πρώτα στον Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσους ε, ε, βοήθησαν στην σύνταξη αυτού του σχεδίου ψηφίσματος και ελπίζω πως ε, θα λάβει μια ευρία υποστήριξη όπως και στα προηγούμενα χρόνια στην Ολομέλεια έτσι ώστε να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ε, προς τους ε, αρμόδιους για τη διαπραγμάτευση. Νομίζω πως αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ στο οποίο αναφέρθηκε και η Πρόεδρος το γεγονό δηλαδή ότι η Συμφωνία των Παρισίων αποτέλεσε μια μεγάλη πρόοδο αλλά οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι εταίροι σε εκείνη τη συμφωνία δεν επαρκούν για την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό είμαι λίγο σκεπτικός όταν κάνουμε αναφορά σε αυτόν τον στόχο τώρα του 1,5 βαθμού Κελσίου, γιατί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ε, επιτείνουμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα και μειώνεται η όθηση που είχε δοθεί με την ε, θέσπιση του στόχου των ε, δύο βαθμών. Και γι' αυτό και στη διάσκεψη στην Βόνη είχα έρθει σε εντατικές επαφέ με τους εταίρους μας από άλλες χώρε του κόσμου, από άλλε περιοχέ του κόσμου και του είχα ρωτήσει ε, ποια είναι η βούληση από τη δική του ε, πλευρά να προβούν σε περαιτέρω δεσμεύσει πέραν δηλαδή των δεσμεύσεων ε, από τη Συμφωνία των Παρισιών. Αλλά για μεγάλη μου απογοήτευση οι περισσότεροι δεν γνώριζαν καν σε τι αναφέρομαι. Δηλαδή μόνο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε στην ανάγκη του να κινηθούμε πέρα από τα όσα συμφωνήθηκαν στη Συμφωνία των Παρισιών. Οπότε ένα πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω προς την Επιτροπή είναι το εξής. Έχει πληροφορίες ως προς το κατά πόσο σε άλλες περιοχές του κόσμου υπάρχει βούληση να αναλυφθούν δεσμεύσεις συμπληρωματικά προς εκείνες που αναλύφθηκαν στην ε, Συμφωνία των Παρισίων. Μετά, στο πλαίσιο της ε, πρόσφατης συζήτησης που κάναμε σε ό,τι αφορά τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είδαμε ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια, δηλαδή να πάμε πάνω από το 40% εάν βρούμε και άλλους εταίρους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν έτσι ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερο τον στόχο των 2 βαθμών Κελσίου. Απλώς όμως δεν βλέπω αυτή τη βούληση και γι' αυτό ρωτάω σχετικά την Επιτροπή αν γνωρίζει κάτι παραπάνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, δομή αν θέλετε εδώ ε, της, ε, του ψηφίσματος, στο σημείο 2 δηλαδή σε ένα σημείο ιδιαίτερα επιφανές αν θέλετε, ε, κάνουμε ε, μία αναφορά η οποία δεν ξέρω αν είναι η καταλληλότερη. Ίσως θα πρέπει να είμαστε ε, από πολιτική άποψη λίγο πιο εμφατικοί, τουλάχιστον στις πρώτες παραγράφους του ψηφίσματος, έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές το ποιοι είναι οι δικοί μας πολιτικοί στόχοι για την επόμενη διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών της κατά την επόμενη κόπη. Επίσης, εδώ γίνεται σαφής αναφορά στον ρόλο των μεταφορών και ευχαριστώ και τον συνάδελφο από το ΕΛΚΕ που έκανε αυτή την πρότασή του να αναφέρουμε δηλαδή την ανάγκη του να υπάρξει μείωση των σχετικών εκπομπών και επίσης γίνεται αναφορά και στο ψήφισμα στην αεροπορία γιατί βέβαια με τη σχετική αδήλωση ξεκίνησε και πρόσφατα μια νέα συζήτηση σε ό,τι αφορά τις εκπομπές της αεροπορίας. Και εδώ απευθύνω έκκληση προς την Επιτροπή αλλά και προς το Συμβούλιο προκειμένου να ε, αποφύγουμε οποιασδήποτε ε, απόπειρε ή οποιασδήποτε εναλλακτικέ προτάσεις προς το Κόρσια, ε, το οποίο ήδη δεν επαρκεί από μόνο του. και ε, ελπίζω η Επιτροπή να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του ε, συστήματος εμπορίας εκπομπών ε, του ETS εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Νομίζω πως αυτή η υποχρέωση βαρύνει και το Συμβούλιο, ότι δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσει θύμα της τωρινής χρονικής συντηρίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Λίζο, κύριο κύριος Λάινα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ε, θεωρώ πως η COP24 θα δείξει τελικά το ποια είναι η δέσμευση την οποία έχουν δείξει και είναι διατεθειμένοι διάφοροι εταίροι να εφαρμόσουν στην πράξη. Δηλαδή θα πρέπει να επιμείνουν στα όσα συμφωνήσαμε τότε στο Παρίσι. Αυτό είναι ο στόχος για το Κατοβίτσε. Και επίσης και εγώ θεωρώ πως έχουμε βρισκόμαστε λίγο πιο μακριά από το στόχο των ε, δύο βαθμών. Και αυτό που θα έλεγα στον συνάδελφο Πεταλίζα είναι ότι οι δύο βαθμοί είναι η υποχρέωσή μας και ο ενάμιση βαθμός είναι ο στόχος. Ε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται και αυτός, αυτή η υποχρέωση εδώ. Δηλαδή, η υποχρέωσή μας να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς, ο στόχος είναι, να, ε, ε, είναι ο 1,5 βαθμός. Ε, και επίση σε ό,τι αφορά την άκρηση πραγματικά ε, ε, και εγώ βλέπω ότι έχει πάρα πολύ σημαντικό είναι μάλλον πολύ χαρακτηριστική σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της καιρικής, των, των καιρικών της κλιματικής μεταβολής. Δηλαδή, ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και ξέρουμε ότι οι θερμοκρασίες έχουν διπλασιαστεί στην Αρκτική σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια ξέρουμε τι θα σήμαινε το λιώσιμο των πάγων. Επίσης, η συμμαχία που έχει δημιουργηθεί ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντική ε, μέσω της ε, ΚΟΠ και βέβαια παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι θα επανέλθουν γιατί βλέπουμε τι έγινε και με την πρόσφατη απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή τα παιδιά κατέληγαν σε φυλακέ των μεταναστών. Τώρα πάλι αποφασίστηκε να υπάρχει επανένωση των οικογενειών. Τώρα υπάρχει και μια τριμερη ε, συνάντηση ε, Κίνα, Καναδά, Κίνας, Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η οποία λαμβάνει χώρα εδώ, σήμερα και αύριο. Οπότε θα ήθελα να μας πει η Επιτροπή τι σκοπεύει να να επιτύχει με αυτή τη συνάντηση για το Πάντω Πάντως ε, σίγουρα δεν επαρκούν οι δράσει μόνο σε κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή χρειαζόμαστε προσπάθειες και σε ε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από τον ιδιωτικό τομέα και από την κοινωνία των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις κύριες πολιτικές, στην εμπορική πολιτική, ε, στην πολιτική μεταφορών και αύριο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα διοργανώσει μια εκδήλωση σε ό,τι αφορά αφορά την κλιματική αλλαγή και τις κρίσεις αλλά ακόμα και τους πολέμους ε, ανά τον κόσμο. Οπότε εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την αποφυγή των σύγκρουσεων. Ε, επίσης αναφέρθηκε πολύ σωστά πως ε, θα πρέπει να έχουμε έναν μακρόχρονο στόχο σε ό,τι αφορά την ε, κλιματική μας ε, πολιτική. Θα πρέπει δηλαδή να αποτελέσει πτυχή όλων των πολιτικών μας και στον σχετικό διάλογο που έγινε στο Βερολίνο πριν από μερικέ μέρες αναφέρθηκε το πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την τις κοινωνικές μεταβολές οι οποίες ε, ε, λαμβάνουν χώρα ως συνέπεια αυτής της ε, αλλαγής. Δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό θα πρέπει να συμβάλλουν όχι μόνο τα διαρθώτικα ταμεία, αλλά και πολλοί άλλοι μηχανισμοί προκειμένου αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού να ολοκληρωθεί σωστά. Μια δηλαδή διαδικασία μεταχειρισμού τόσο ε, περιβαλλοντική όσο και κοινωνική. Και θα υποβάλουμε και κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπαν και ο Πίτερ και ο Τζο. Υπάρχει ένα στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω επίσης. Συχνά μιλάμε για τους στόχους του Παρισιού εγώ έχω διαφορετική άποψη. Πιστεύω ότι το όριο των δύο βαθμών Κελσίου, έτσι το λέω όριο, είναι η γραμμή που δεν πρέπει να υπερβούμε. Είναι το μη παρέκει. Όσο πιο μακριά μείνουμε από τους ε, δύο βαθμούς Κελσίου, τόσο το καλύτερο. Λιγότερες συνέπειες θα έχουμε, λιγότερη κλιματική αλλαγή θα δούμε. Όσο πιο κοντά πλησιάσουμε στο 1,5 βαθμό Κελσίου, τόσο το καλύτερο. Δεν νομίζω ότι αν τονίσουμε λοιπόν το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου δεν θα, θα, θα απογοητευτεί ο κόσμος. Αντίθετα θα τον βοηθήσουμε να καταλάβει πόσο κατεπήγον είναι το πρόβλημα και πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Γιατί ο χρόνος που έχουμε για να μην ξεπεράσουμε την αύξηση του 1,5%, του 1,5 βαθμού Κελσίου είναι πολύ λίγος. Και μια και οριστικοποίησαμε τις μεγάλες διαπραγματεύσεις ε, για την ενέργεια με το Συμβούλιο αυτή τη βδομάδα και αυτό οδήγησε στην παρατήρηση του Επιτρόπου Κανιέτε ότι τώρα μπορούμε να αυξήσουμε τις εθνικές προθέσεις συνεισφοράς ε, στο 45%. Το 40%. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ε, κίνηση που κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης IPPC ότι θέλουμε να αυξήσουμε τις δικές μας συνεισφορές σε σχέση με τις συνεισφορέ που κάναμε στο Παρίσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και παράλληλα αισθάνομαι μια ελαφρά απογοήτευση, για να μην πω ισχυρή απογοήτευση, για τη γενική στάση των κρατών μελών σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το σύστημα εμπορίας εκπομπών, για τον καονισμό, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και για όλους τους φακέλους της ενέργειας που είναι πάρα πολύ μινιμαλιστικοί. Δεν θέλουμε, είναι σαν να μην θέλουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και να στηρίξουν την αγώνα. Η στάση είναι γενικά... Ποιο είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε έτσι για να ξεπετάξουμε το θέμα. Και αυτό οδηγεί όχι μόνο σε μη φιλόδοξους στόχους, αλλά οδηγεί και σε έλλειψη ενός ε, νομικά δεσμευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Μοιάζει τα κράτη-μέλη να μην είναι έτοιμα, διατεθειμένα να δεχτούν νομικά δεσμευτικές ε, συνεισφορές ε, ούτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση πολλό δε μάλλον σε επίπεδο εθνικό. Ε, παρότι κάνανε πολλές προσπάθειες αποτελεσματικέ αποτελεσματικές μέχρι τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δύο τελικές παρατηρήσει, αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε. Καταρχάς, η στρατηγική για το 2050 είναι πάρα πολύ σημαντική και καλό ακόμα μια φορά τα κράτη-μέλη να μην θεωρήσουν ότι είναι ασήμαντη αυτή η στρατηγική. Θα οδηγήσει στον εξή στόχο να έχουμε μηδενικές εκπομπές το 2050 και να περάσουμε και σε αρνητικές εκπομπές μετά το 50. Ελπίζω τελικά τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να δεσμευτούν, γιατί δεν ήταν όταν συζητήσαμε το φάκελο για τη διακυβέρνηση της ενέργειας. Και ελπίζω ως Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε σε θέση να έχουμε ε, ισχυρότερες δεσμεύσεις για το Διεθνές Σύστημα Χρηματοδότησης. Δεν έχουμε ένα αυτόματο σύστημα όπου τροφοδοτούμε το Ταμείο για, την, ε, για το κλίμα. Και αν θέλουμε πραγματική κλιματική διπλωματία και αν θέλουμε να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο ότι πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, καθώς και τις, ε, ανα, τις υπόλοιπες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τότε θα πρέπει να δεσμευτούμε πολύ περισσότερο και να προσφέρουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Ο κ. Σέικχαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συντάκτες του, του ψηφίσματος. Το ψήφισμα αυτό πιστεύω είναι μια καλή βάση για τη συζήτηση και αργότερα στην Ολομέλεια. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι η συνάντηση στο Κατοβίτσε, το COP24, θα είναι πολύ κρίσιμη. Είναι η χρονιά της αναθεώρησης πριν αρχίσει πραγματικά να ισχύει η Συμφωνία του Παρισιού. Είναι η χρονιά όπου και οι διεθνείς εταίροι δεσμεύτηκαν να αντιδράσουν στην έκθεση IPPC για τον 1,5 βαθμό Κελσίου, έκθεση που θα δημοσιευθεί αρχές Οκτωβρίου. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα επιτάπητος και νομίζω ότι θα είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση COP. Ε, και καλό είναι να είναι έτοιμη η Ευρώπη, να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και αυτό, αυτό δίνει Ω μήνυμα και το ψήφισμα. Ε, Μία-δύο ερωτήσει προ την Κομισιόν. Καλή είναι η χρονική στιγμή, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντική και για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει του επόμενου έξι μήνε, γιατί ακολουθούν μια σειρά από συνεδριάσει. Λοιπόν, αυτό που θέλω να μου πει η Επιτροπή είναι τι προβλέπει ε, για την Ευρώπη. Πώς θα αυξήσει η Ευρώπη τις δικές της προθέσεις ε, συνεισφοράς. Ε, γιατί ο κ. Κανιέται είπε ότι μπορούμε να πάμε από το 40 στο 45. Θα προταθεί αυτό επίσημα, η είναι απλώς μια δήλωση του Κανιέται που είναι έτσι για εσωτερική κατανάλωση. Θα δούμε επίσημη πρόταση. Υπάρχουν ε, συνεδριάσεις στην Πανκόκα, από ό,τι ξέρουμε και στις αρχές του Οκτωβρίου ε, θα υπάρχει η έκθεση για τον 1,5 βαθμό Κελσίου και Πίτερ ε, Λίσε. Εμείς μιλάμε για ένα όριο για να μείνουμε πολύ κατά, πολύ πίσω από τους δύο βαθμούς Κελσίου ε, και κατά προτίμηση στο 1,5, στο 1,5 βαθμό. Ε, αυτό θέλουμε. Υπάρχει στη Συμφωνία του Παρισιού, την επικυρώσαμε όλοι. Αυτό είναι ε, που αυτό πρέπει να κάνουμε, να μείνουμε πολύ πιο κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου και αν μπορούμε και κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου. Και στην έκθεση του IPPC τον, τον Οκτώβριο, αυτό που θα δούμε είναι ότι οι επιπτώσεις ε, της ε, κλιματικής αλλαγής είναι τελείως ε, διαφορετικές ανάλογα με το στόχο του 2 ή του 1,5 βαθμού Κελσίου. Αν περάσουμε το 1,5 στους 2 βαθμούς Κελσίου θα είναι πολύ διαφορετικές οι επιπτώσεις και πρέπει να την κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Νομίζω λοιπόν και εξώ και το ερώτημα στην Κομισιόν ότι πρέπει να μου πείτε ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ετοιμάζεται ένα οδικό χάρτη για τον Νοέμβριο, για το 2050. Θα συνδέσετε εκεί, α, το, εκεί θα μιλήσετε και για το στόχο του 1,5 βαθμού. Ε, αυτό σημαίνει υψηλότερου στόχου, υψηλότερε φιλοδοξίε. Το ζητάνε ένα-δύο, μια-δύο χώρε. Α πούμε, Μέχρι το 2030 η Ολλανδία ζητάει μείον 55%. Αυτή την ε, εβδομάδα ο, η Μέρκελ και ο Μακχό συναντιούνται και θα κάνουν κοινή ε, δήλωση. Θα πούνε για την Ευρωζώνη και τους ε, πρόσφυγες, αλλά θα πούν ότι η Ευρώπη θέλει να, πρέπει να αυξήσει τις φιλοδοξίες της στο COP24. Πώς θα εξασφαλίσει η Κομισιόν ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι, ούτω ώστε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχουν σημασία. Περιμένω λοιπόν την Κομισιόν να μου ξεκαθαρίσει λίγα και το τοπίο, για πώς βλέπετε να ε, ετοιμαστούμε τον, ε, το επόμενο εξάμεινο με προοπτική το Κατοβίτσε. Τώρα για την, για την ε, αεροπορία. Μιλάμε για την εφαρμογή του Κορσία. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κρατήσει το δικό της σύστημα εμπορίας εκπομπών. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η Κομισιόν αλλά και όλα τα κράτη-μέλη θα κάνουν επιφύλαξη εάν το Κορσία ε, κινηθεί προς την κατεύθυνση που μοιάζει να κινείται τώρα. Δηλαδή ότι είναι για όλες τις ε, διεθνείς ε, πτήσεις. Και ξέρω από την ότι οι διεθνείς πτήσεις είναι και οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις. Και αυτό δεν θα πρέπει ποτέ να το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κορσία. Και θέλω να μου το πείτε ξεκάθαρα. Θέλω να μου το πει ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού θα εξασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζουν κάτι τέτοιο ε, καθώς εκπονείται περαιτέρω με το Κορσία ε, στα πλαίσια της ΕΚΑΟ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και το θέμα του Κορσία βεβαίως που θα συμπεριλάβουμε στη συζήτηση και θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει κατόπιν του αιτήματός μας. Τώρα έχουμε Έχω και άλλους συνεισηγητές στον κατάλογο, αλλά δεν είναι εδώ. Επομένως, ε, θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ε, βουλευτές. Η κυρία Κονέτσινα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της ε, σκιώδης ηγητριάς μας, της Στεφάνια Τόρες, η οποία δεν θα μπορέσει να είναι εδώ σήμερα και ζητά συγγνώμη. Θα διαβάσω κάποια από τα σχόλιά της. Το σχέδιο ψηφίσματος για την COP24 αναγνωρίζει τα επιτέχματα των COP22 και COP23 και περιμένει ότι τα αποτελέσματα ε, του 2018 θα παρουσιαστούν ε, στην COP24. Πρόκειται για μια παγκόσμια διαδικασία επικοδομητικής συζήτησης και λύσεων που προτείνονται από τις κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακαδημαϊκό τομέα, επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ότι ε, η ε, ισχύς ε, της ενέργειας είναι καθοριστικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό και δεν θα έχουμε καμία πρόοδο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Στη διάρκεια της COP24 είναι πολύ σημαντικό να επιμένουμε στο ρόλο των γυναικών και στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πέρσι ε, εγκρίθηκε το πρώτο γενικό σχέδιο. Υπάρχει όμως το πρόβλημα ότι το συμφωνημένο σχέδιο δεν υπάρχει, δεν αναγνώρισε την ανάγκη να αναφερθούν οι γυναίκες, ε, οι ακτιβιστές υπέρ ε, των θεμάτων αυτών και επίσης πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους ενεργειακούς πόρους και να συμπεριληφθούν οι γυναίκες, διότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα αιτήματα τα οποία παραβλέφθηκαν στην COP23. Υπάρχουν αρκετέ οργανώσει στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία που οργάνωσαν ε, κινήσει για τα θέματα αυτά και η εκπροσώπηση των γυναικών και των ανθρώπων που υπερασπίζονται το κλίμα ήταν ελάχιστη. Άρα το πρόβλημα είναι συστημικό. Χρειαζόμαστε γενικότερη αλλαγή στο οικονομικό σύστημα και στον τρόπο ζωής μας. Στη διάρκεια της COP23 η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις εκπομπές επετέφθη επιτέλους και σχεδιάζεται για το 2020 μετά από την κύρωση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας ε, των αλλαγών της Ντόχα, που είναι η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιώτο 2013-2020 και ε, τη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σχέση με το 1990. Αλλά αυτά ήταν τα ελάχιστα. Αυτό που χρειαζόταν στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο επίπεδο φιλοδοξίας, ε, αλλά ε, ως συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε τα πάντα για του χρόνου. Θα επαναλάβουμε το ίδιο σενάριο λοιπόν ε, δεσμεύσεων ε, στην Κατοβίτσε και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα από μία σύνοδος για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και ε, φυσικά δεν ε, ε, δίνεται η μάχη στα θεσμικά όργανα. Χρειαζόμαστε στους ανθρώπους στους δρόμους αλλά και στα σπίτια τους σε καθημερινή βάση να δίνουν μάχη για ε, την καταπολέμηση της φτώχειας, να υπάρχει ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη. Η πόλη είναι σημαντικός παράγων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι πόλεις όπως για παράδειγμα πόλεις μεγάλες όπως η Βαρκελόνη, δίνουν το παράδειγμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά στην COP24. Οι πόλεις πρέπει να συμμετέχουν στις ε, αποφάσεις, πρέπει να ακούσουμε τα αιτήματά τους, διότι ε, χρειάζονται αυτονομία, υποστήριξη και χρηματοδότηση. Για να καταπολεμήσουμε λοιπόν την κλιματική αλλαγή και να κάνουμε αλλαγές για να μετριάσουμε τις αλλαγές, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συμφωνίες ε, που να μην πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση από την κυριαρχία των τροφίμων και μιας διαφοροποιημένης τοπικής οικονομίας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια άσκηση ειλικρίνειας στον τομέα αυτό. Και εν τέλει πιστεύω ότι θέλω να πω ότι... Ε, ευχαριστώ πολύ διότι είχαμε ένα πρώτο θετικό βήμα εχθές στην ψηφοφορία με την έγκριση ενός κοινού ψηφίσματος με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και θέλουμε να ευχαριστώσουμε όλους εκείνους που συμμετείχαν διότι ε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και για το μελλοντικό μας έργο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άντριο Κούπερ, ο οποίος είναι εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Κούπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Καλωσορίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος ε, της ε, MV για την COP24, καθώς επίσης και την έγκριση της έκθεσης για τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις ε, για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Τονίζουμε το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε αυτή την έκθεση και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή του 70% των μέτρων μείωσης των συνεπειών του κλίματος και ε, μέτρων προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος. Ε, όταν λοιπόν οι κυβερνήσεις νομοθετούν, οι πόλεις και οι περιφέρειες αναλαμβάνουν τα ενία. Ε, υπάρχει λοιπόν αυξημένη ευθύνη για τις τοπικές κυβερνήσεις και ε, τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Αυτό τονίστηκε και πέρσι στη Βόνη, στην έναρξη ε, του κοινού διαλόγου και των δεσμεύσεων της ε, Βόνης. Πρέπει λοιπόν αυτή η μορφή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης να αναγνωριστεί πλέον και ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών να επισημοποιηθεί ως τμήμα της διακυβέρνησης της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος. Η πρόσφατη στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση κυβέρνηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνία του Κλίματος. Χωρίς κατάλληλη σύμπραξη μεταξύ τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων, θα είναι ακόμα δύσκολο να επιτύχουμε και αυτού του στόχους θα πρέπει να μειώσουμε την αύξηση κατά 2% και αυτό, 2 βαθμούς, συγγνώμη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα, χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα έχει τοπικές και περιφερειακές ε, ε, διαδικασίες ε, συμβολής, οι οποίες θα συμπληρώσουν την εθνική προσπάθεια. Τα περισσότερα γίνονται σε τοπικό επίπεδο και ξέρουμε ότι οι δράσει οι οποίε δεν προσμετρούνται, ούτε αναγνωρίζονται, ούτε ενθαρρύνονται, ούτε αξιολογούνται. Επομένω, αυτέ οι τοπικέ δράσει ε, που θα μπορούσαν να είναι πιο σημαντικέ, ε, είναι αυτέ οι οποίε θα κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιτυχία και αποτυχία. Γι' αυτό ακριβώ και ζητούμε ένα πλαίσιο διαφάνεια, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει εθνικέ εκθέσει ε, που θα έχουν μια ειδική ενότητα αφιερωμένη σε επίπεδα κάτω του εθνικού γενικού επίπεδου ε, για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους. Ο διάλογος φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικός για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, διότι μας επιτρέπει να προωθήσουμε τις φιλοδοξίες μας, τις θέσεις μας και τις προθέσεις μας και φυσικά θα πρέπει να ε, δίνουμε και στοιχεία για την εφαρμογή των δράσεων για το κλίμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαμορφώσουμε τι μελλοντικέ ε, πρωτοβουλίε πολιτική. Ο διάλογο δεν θα πρέπει να είναι μονόλογο. χρειαζόμαστε διτή επικοινωνία, πρέπει να εισακουγόμαστε, αλλά πρέπει να μα απαντούν κιόλα. Επίση πρέπει να συμπεριλάβουμε τα αποτελέσματα του διαλόγου στο κείμενο τη διαπραγματεύση τη ΚΟΠ και ε, θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνεται και στην ΚΟΠ 24. Η συνεργασία και η συμπερίληψη όλων αυτών των στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να έρθουν σε επαφή με τι δημοκρατικέ ε, εκκλησμένε τοπικέ αρχέ και περιφερειακέ αρχέ και φυσικά την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Και πρέπει φυσικά να μιλάμε με μία ενιαία φωνή στην COP24. ω ερετά μέλη τη πιο κοντινή κοινότητα των πολιτών θέλουμε να βοηθήσουμε να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Τέλος, ως μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου της Επιτροπής των Περιφερειών, γνωρίζω σαφέστατα ότι το Brexit, ή ελπίζω τουλάχιστον να μην υπάρξει Brexit, ακόμα ελπίζω, ελπίζουμε να μειώσουμε και του στόχους της, μείωση μείωσης χρήση χρήσης του άνθρακα, διότι πραγματικά θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην υστερήσει περαιτέρω στις δράσεις του το Ηνωμένο Βασίλειο αν είναι μόνο του δεν θα μπορεί να συγκρίνει την πρόοδό του. Μαζί σας έχουμε καλύτερες πιθανότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε από τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Δύο μιλητές ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να είστε σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Γιατί έχουμε και τον ε, ψήφι μας που μας περιμένει έξω από την αίθουσα για το επόμενο σημείο. Κύριε Βυζινιέστηκα λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πραγματικά χαίρομαι για το γεγονό ε, που θα λάβει χώρα στο ε, Κάτοβιτς η φετινή κόπ. Ελπίζω να είστε όλοι εκεί και να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της διάσκεψης. καθώς βέβαια στόχος κοινός εκεί είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, προφανώς οι στόχοι που τέθηκαν στην Συμφωνία των Παρισίων ε, είναι ένα κοινό μας επίτευγμα, αλλά πώς θα καταφέραμε τελικά να ορίσουμε αυτούς τους στόχους, ε, αποφεύγοντας ε, την μείωση των εκπομπών του άνθρακα γενικά, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις, ε, την αναφορά στις σχετικές καλλιέργειες και το ρόλο που παίζουν στις εκπομπές ε, άνθρακα. είχε γίνει είχαν γίνει σημαντικές αναφορές σε σχέση με αυτό το ζήτημα από τη δική μας ε, πλευρά, από τη δική μου χώρα και το αρμόδιο Υπουργείο και βλέπουμε τώρα πως τελικά φτάνουμε σε ένα σχέδιο ψηφίσματος όπου ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για, μια, για ένα κλάδο εδώ μηδενικών εκπομπών κατά τη δική μου άποψη είναι αμφίβολο το κατά πόσο θα μπορούσε να ε, εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην πράξη. Και το επαναλαμβάνω εδώ, η Συμφωνία των Παρισίων κατέστη δυνατή όταν διαγράφηκε από αυτή η μείωση των εκπομπών άνθρακα, το decarbonization. Και ε, όταν κάνουμε λόγο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτήν την, ε, τις μηδενικές εκπομπές, ε, τότε αυτό δεν επαρκεί, γιατί εμείς ε, σήμερα είμαστε υπεύθυνοι για το 10% των παγκοσμίων εκπομπών. Οπότε το να κάνουμε εμείς μια προσπάθεια μονομερός δεν έχει καμία σημασία. Και κάτι ακόμα που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί ένας τέτοιος στόχος χωρίς τεράστιο και οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, ε, συμπεριλαμβανομένες της ε, και γενικότερα της Πολωνίας. Ε, πάντως σε κάθε περίπτωση σας ε, περιμένουμε στο Κατοβέτσε και ακριβώ ε, προκειμένου να διατηρήσω το πνεύμα τη Συμφωνία των Παρισιών, θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε έτσι ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα αφενός ε, στη μείωση των εκπομπών και από την άλλη και αφετέρου ε, την ε, δέσμευση αυτή, την αποθήκευση αυτών των εκπομπών. Και ένα τελευταίο σχόλιο να πω ότι η επόμενη λοιπόν διάσκεψη κορυφής θα λάβει χώρα στο Κατοβίτσα. Το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει με τις διαπραγματεύσει που είχαν γίνει σε ό,τι αφορά την Ενεργειακή Ένωση και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να δώσουμε την πλήρη υποστήριξή μας σε αυτή τη διάσκεψη. Σας ευχαριστώ πολύ. επειδή έχουμε τον ομιλητή ο οποίος ήδη μας ε, περιμένει για το επόμενο σημείο της σημερινής σας διάταξης, θα δώσω άμεσα τον ε, κύριο Μέντους. Ε, και ζητώ συγγνώμη στου ε, υπόλοιπου συναδέλφου. Και η κυρία Γούτελαν, για παράδειγμα, ζήτησε το λόγο, αλλά δεν μπορώ να τη ε, την δώσω. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή έχει το λόγο ναι, ευχαριστώ να πω ότι καταρχήν χαιρετίζουμε αυτό το ψήφισμα από την πλευρά τη Επιτροπή σα σε ό,τι αφορά το Κατοβίτσε. Ε, νομίζω ε, πως ε, από την έκθεση της IPCC ένα 5, πως χρειάζεται να αναλυφθεί δράση από την πλευρά όλων προκειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έχουμε όχι μόνο τον κανονισμό για τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή που δημοσιεύτηκε, ε, που περιλαμβάνει και την ε, μεταρρύθμιση του ETS, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε και τις ε, διάφορες νέες διατάξεις για την διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Και πραγματικά αυτό είναι θετικό, ότι βλέπουμε δηλαδή νομοθετικά να απηχείται αυτό αυτή η βούλησή μα και ε, επιχαίρουμε επίση το γεγονό ότι σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό σταθεροποίηση τη αγορά, απέρριψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σήμερα μια σχετική προσφυγή. Ε, εμείς συνεχίζουμε τι προσπάθειε μα, Ο κύριο Κανιέτη συμμετέχει σήμερα στην Υπουργική Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή συνομιλώντα με του συναδέλφου μα από την Κίνα αλλά και από τον Καναδά οι οποίοι από τη δική του πλευρά διαμορφώνουν το δικό του σύστημα τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα με βάση το δικό μα πρότυπο, το ευρωπαϊκό. Αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω δράση σε διάφορα επίπεδα. Ο Επίτροπος Κανιέται συνεργάζεται με τον Καναδά, την Κίνα και την συμμαχία υψηλή φιλοδοξία, ειδικότερα τι χώρε του Ειρηνικού. Και όπω αναφέρθηκε ήδη από τον συνάδελφο, αύριο θα λάβει η χώρα μια σημαντική συνάντηση ε, με την ε, πρόεδρο ε, Μογκερίνη, με διάφορου υπουργού εξωτερικών. Ε, και ο δικό μα ε, Γενικό Διευθυντή βρέθηκε πρόσφατα στην Κίνα, όπου προβήκαμε σε μια ανταλλαγή εμπειριών σε ό,τι αφορά τι δράσει που αναλαμβάνουμε για τη μετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει όσα μπορεί, οι υπόλοιπε περιοχέ θα πρέπει να κάνουν κι άλλα και τι βοηθάμε σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα στοιχεία που μα αφορά στην ΚΟΠ. Ε, ένα άλλο στοιχείο είναι βέβαια η οριστικοποίηση τη λίστα των κανόνων από την ΚΟΠ των Παρισιών, έτσι ώστε να υπάρχουν κοινοί κανόνε σε ό,τι αφορά την ανάληψη των ευθυνών, τη διαφάνεια και αλλά και προκειμένου οι διάφορες ε, δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν ε, να έχουν ε, και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Τώρα αναφέρθηκε η μεσοπρόθεσμη στρατηγική και αν δούμε την την έκθεση ε, σε ό,τι αφορά τον 1,5 βαθμό. Ε, πράγματι υπάρχουν μεγάλες ε, ομοιότητες εδώ ανάμεσα στα όσα εμεί προτείνουμε και τα όσα αναφέρει η έκθεση και σε επίπεδο πόλεων, δήμων και κοινοτήτων. Γιατί πραγματικά χωρίς τη συμβολή όλων αυτών των φορέων δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον στόχο του 1,5 βαθμού. Και εδώ χρειαζόμαστε δηλαδή μια συλλογική φιλοδοξία. Η Επιτροπή δηλαδή επιθυμεί να υπάρξει μια γενικότερη συλλογική βούληση προκειμένου να αυξήσουμε όλες τις καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς. Ε, και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε ο, ο κύριος ε, ε, ε, Πεταλίζε σε ό,τι αφορά την, ε, τονικά. ε, και πράγματι εδώ θα προβούμε σε μια σχετική ενημέρωση και των κρατών από την πλευρά τη Επιτροπή. Όλα δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό. Και για το Κοινοβούλιο υπήρξε σαφέ σε σχέση με αυτό το ζήτημα εδώ και σειρά ετών. Ω προ το τι θα συμβεί, μπορώ να σα πω το εξή. Στο παρελθόν, όταν ε, ε υιοθετούμε ε, διεθνείς διατάξεις και υπάρχει διαφορά με το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, υπήρξαν ε, διαδικαστικές διαφορές ε, προκειμένου να αλλάξει η η νομοθεσία εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εξωτερικέ συμφωνίε δεν μπορούν να μεταβάλουν την ενωσιακή νομοθεσία χωρί τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ε, Τέλο, σε ό,τι αφορά τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς ε, και την αναφορά που έγινε σε ό,τι αφορά τη χθεσινή δήλωση ότι δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε σε ε, μείωση κατά 45% με βάση τις ε, προθέσεις συνεισφοράς που έχουμε σήμερα. Ναι, αυτή είναι η πρόθεση και δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε κάτι διαφορετικό στα Ηνωμένα Έθνη στο εγγύς μέλλον, απλώς αναφέρθηκε από τον Επίτροπο χθε το τι σκοπεύουμε να κάνουμε, ποιος είναι ο στόχος μας. Και όπως και στο προηγούμενο σημείο ε, της παρέμβασής μου, ε, το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο ε, συμμετέχουν ενεργά στο πλαίσιο της όλης αυτής της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Not for good because... Με τη συζήτηση για το COP24, καλώς ορίζω τον προσκεκλημένο μας, τον δόκτορα Σολχάιμ, εκτελεκτικό διευθυντή του περιβαλλοντικού προγράμματος του ΟΗΕ Εδώ και δύο χρόνια είσαστε επικεφαλής του UNEP. Μετά την υιοθέτηση ακριβώς της Συμφωνίας του Παρισιού αναλάβατε τα ενία. Δεδομένης της σημασίας του οργανισμού σας, ε, δεδομένου του διακυβεύματος ε, της καταπολέμησης, δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, η Επιτροπή μας προσπαθούσε πάντα να διατηρεί στενές ε, σχέσεις και συνεργασία με τον οργανισμό σας στα πλαίσια της ετήσιας Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα ε, έχετε συναντηθεί με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω και στο, στη συνάντηση υψηλού επίπεδου ε, τον Ιούλιο και αργότερα στην COP24 στο Κάτοβιτσε να ξανασυναντηθούμε ε, γιατί να καταλάβουμε την άποψη φορέων όπως του UNDP για τις εξελίξεις στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής. Ο διάλογος της Ταλανοά ε, συμφωνήθηκε στο COP23 και είναι να εξελίξει με κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα που θα προκύψουν στο τέλος του 2018. Ε, περιμένουμε και τη δημοσίευση της έκθεσης του IPPC για τον, τον 1,5 βαθμό Κελσίου ε, το φθινόπωρο η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι τεράστιο θέμα ε, και το άλλο θέμα είναι ε, η μετάβαση σε μια παγκόσμια κυκλική οικονομία και όλα αυτά που συνεπιφέρει. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας λοιπόν για αυτά τα θέματα και σας δίνω το λόγο ακριβώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ούτε την κλιματική αλλαγή, ούτε κανένα άλλο μείζον θέμα του πλανήτη. Ξέρετε ποιος είμαι, αλλά ας το επαναλάβω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην καρδιά αυτού που θέλουμε να πετύχουμε και ο ΙΕ και αντιμετωπίζουμε μαζί κοινέ προκλήσεις. Πρέπει να αλλάξουμε φυσικά το αφήγημά μας, να πούμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά όπω και να έχει το πράγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στον πυρήνα τη προσπάθεια. Χωρί αυτή δεν γίνεται. Ε, υπάρχουν βεβαίω ε, πιθανοί σύμμαχοι, μεγάλοι σύμμαχοι όπω η Κίνα, για να πετύχετε αυτό που θέλετε. Την ξέρετε την ε, κατάσταση. Έχουμε αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα δεδομένα για την ανθρώπινη ιστορία. Ε, Δίνουμε περισσότερη ε, ηλιακή ενέργεια στο παγκόσμιο δίκτυο από οποιαδήποτε ενέργεια που παίρνουμε από το φυσικό αέριο κτλ. Ε, δεν θέλω να σας μιλήσω για την τεράστια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Τα ξέρετε όλα αυτά. Και αν δεν ξέρετε κάτι, ε, μπορώ να το διευκρινίσω αργότερα. Αλλά ας περάσουμε τώρα στην καρδιά της συζήτησης. Η πιο συχνή ερώτηση που μου κάνω όταν ταξιδεύω είναι τι θα γίνει με τον Donald Τραμπ. Είναι λιγότερο σημαντικό για το κλίμα και το περιβάλλον από ό,τι νομίζουμε όλοι μας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα σεβαστούν κατά πάσα πιθανότητα την Συμφωνία του Παρισιού λόγω της οικονομικής συγκυρίας ε, λόγω του οικονομικού αμερικανικού μοντέλου, Microsoft κτλ. Όλοι πιστεύουν, όλες οι μεγάλες εταιρείε πιστεύουν ότι χρειάζεται κάποια δράση για την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή. Μπορεί να είναι πιο αργή από εμά, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι το νέο μοντέλο οικονομίας και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έχουν, δημιουργούν πενταπλάσια πενταπλάσιες θέσεις απασχόλησης ε, από την στον τομέα της παραγωγή ηλιακή ενέργειας από ότι στον τομέα του άνθρακα, χάλιβα και τι παραδοσιακέ ε, βιομηχανίε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ε, θα κατέβουν ξανά στην, ε, στο πλανήτη Γη. στο Κεντάκι όταν φτάσανε πρόσφατα, γιατί μιλήσανε στην πραγματικότητα, πάλι για την ηλιακή ενέργεια στην Αμερική. Και αυτό ακριβώς συμβολίζει τη δύναμη της ηλιακής ενέργειας, ε, που είναι φοβερά ανταγωνιστική. Όλοι ξέραμε και για το ότι ήταν καλό, καλή η ηλιακή ενέργεια και για το περιβάλλον και για την υγεία. Είναι καθαρή ενέργεια, αλλά είναι ακόμα καλύτερη γιατί είναι και φθηνή ενέργεια. Και αυτό ε, είναι σημαντικό γιατί το συνειδητοποιούμε τώρα και διάφορε οργανώσει κοινωνία των πολιτών, διάφορε πολιτείε όπω η Καλιφόρνια και ο ιδιωτικό τομέα θα πιέσουν το ομοσπονδιακό επίπεδο των... και την κυβέρνηση των Αμερικανών να σεβαστεί τι ε, δεσμεύσει του Παρισιού. Η Ευρώπη έχει σημαντικότερου ε, συμμάχους πέρα από αυτού. Η Κίνα αλλάζει ε, τη στάση της για το περιβάλλον. Μπορείτε να μην υποστηρίζει την Ευρώπη 100%, αλλά κινείται με μια ταχύτητα ανεκδίγητη ε, και ε, τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος ε, ενδιαφέρονται και υπόθηκε στο συνέδριο του Εθνικού Κομμουνιστικού Κόμματος ότι το επόμενο ε, πενταετές πλαίσιο θα έχει ε, να κάνει με τα θέματα της ενέργειας και την ελάφρυνση της φτώχειας. Ε, και ακριβώς γιατί επειδή έχουν αλλάξει στο Πεκίνο τα τελευταια τρια 3-4 χρόνια η μολις εχει έχει μειωθεί κατά 30-40%. Ε, προστασία του νερού, ε, καθαρισμός των ποταμών, κάνουν τεράστιες προσπάθειες με τεράστια ταχύτητα, ε, που τα κάνουμε εμείς στην Ευρώπη, αλλά στην Κίνα τα κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Ας χαιρετήσουμε αυτή την πρόοδο. Ε, επομένως, η Κίνα και η Ινδία ε, είναι φυσικοί σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και το καλύτερο δεν το κάνουν για μας, για μας τους Ευρωπαίους, το κάνουν για τον εαυτό τους. Πριν από 10 χρόνια, από το 2007 και μετά, κάναμε διάφορες συζητήσεις ε, και η Ευρώπη ε, σκεφτόταν ότι έπρεπε να, πιστε... να πείσει τους Κινέζους να κάνουν κάτι για το κλίμα. Ε, ότι ήταν σημαντικό για τον κόσμο, δεν το καταλαβαίνανε, αλλά έπρεπε να τους πείσουμε. Μετά ο Ντόναλτ Τραμπ έβγαλε τις Ηνωμένε Πολιτείες από τη συμφωνία του Παρισιού. Οι Κινέζοι τι είπανε. Ότι αν δεν κάνουμε κάτι για το κλίμα ε, και δεν κάνουμε κάτι τώρα θα είναι έγκλημα για τις επόμενες ε, γενιές. Και η Ινδία το είπε αυτό. Αυτό είναι τεράστια διαφορά η Κίνα και η Ινδία λοιπόν γίνονται φυσικοί μας σύμμαχοι ε, στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Πάμε λοιπόν για τις συζητήσεις στο Κατοβίτσε, στην Ευρώπη. Επομένω, έχει την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια. Ε, οι κοδεσπότε είναι οι Πολωνοί. Είναι τεράστια η σημασία τη εκδήλωση. Ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε για την ανακοίνωση αυτή και τα θέματα που θα προκύψουν, αλλά τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ε, πιο ευρεία εικόνα. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το κείμενο το οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς ε, στις διαπραγματεύσεις. Πιστεύω και το έχω συζητήσει με διάφορους ε, επιτρόπους στις Βρυξέλλες ότι πρέπει να αλλάξουμε το αφήγημα. Μιλούσαμε για το κλίμα, το οποίο ήταν πιστικό για πολλούς αλλά δεν μπορέσαμε να το κάνουμε καθημερινή συζήτηση για όλους τους λαούς. Ο κόσμος δεν το συζητάει, δεν συζητάει το κλίμα. Είτε στο Γκουαντόγκ ε, συναντιούνται οι αρχηγοί, είτε ε, στη Γλασκόβη, είτε στο Τωρίνο, είτε οπουδήποτε. Γιατί, γιατί μερικέ φορέ είναι δύσκολη αυτή η γλώσσα. Ε, δεν μπορεί ο κόσμο να καταλάβει αυτά τα θέματα. Ε, θα πρέπει να το κάνουμε. Κάποιο είπε, Αμερικάνος, ε, αν πάω στην Αϊόβα ε, και πω ας πούμε ότι θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας α πούμε στη Φλόριδα, δεν δίνουν διάρα οι κάτοικοι της Αϊόβα. Ε, θα πρέπει να πιστούν πώς θα τους επηρεάσει τους ίδιους. Γιατί κάτι τέτοιο θα τους πείσει. Να μιλήσουμε μια γλώσσα που θα τους, ε, που τους να αποφύγουμε τα τεχνικά κρονίμια, τα οποία είναι τα βλέπουμε παντού σε όλε τι ανακοινώσει. θα πρέπει την κλιματική αλλαγή και τον αγώνα κατά τη κλιματική αλλαγή να την συνδέσουμε με οικονομικέ ευκαιρίε, δημιουργία θέσεων απασχόληση. ε, περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, στο τομέα τη ηλιακή ενέργεια, από ό,τι στον Νάθακα και χάλιβα και για τι γυναίκε, καλύτερε θέσει απασχόληση, με καλύτερου μισθού, Να συνδέσουμε λοιπόν την, τον αγώνα αυτό με την οικονομική ευημερία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Αυτό κάνουν διάφοροι πρωθυπουργοί και στην ε, ε, Κίνα και στην, και ε, στην Ινδία. Ε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντλίες, να αντλήσουμε ενέργεια για να έχουμε καθαρότερη ενέργεια σε διάφορα μέρη της Ινδίας στον, και της Κίνας, στον τα κτλ. Και αυτό θα είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους και για τις γυναίκες κτλ. Τώρα λοιπόν ε, μπορούμε επίση να δώσουμε ενέργεια, φθηνή ενέργεια σε χωριά και σε πόλεις που δεν είναι συνδεδεμένες ας πούμε, στην ιδέα με το δίκτυο. Ε, να πείσουμε τον κόσμο ότι αν θα το κάνει, ε, αν δεν χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για το καλό του ε, κλίματος, να το κάνει τουλάχιστον για την οικονομία. Ε, είναι καλό για όλους αυτό, είναι καλό για τους ε, μετόχους, για τις θέσεις απασχόλησης, για το περιβάλλον, για την οικονομία. Πρέπει να περάσουμε στην ηλιακή ενέργεια λοιπόν. Να αλλάξουμε λοιπόν επίσης τη γλώσσα. Να υπάρχουν και στενότεροι δεσμοί με την οικονομία και να περάσουμε στα θετικά. Μπορώ να τα καταφέρω, διότι πολλοί συζητήσεις για το κλίμα είναι αρνητικές και αναφέρονται στις αρνητικές συνέπειες της αδράνειας. Και φυσικά αυτό είναι τρομακτικό. Αν αδρανήσει κανεί, θα έχουμε περισσότερε πλημμύρε, ξηρασία, θα αυξάνει το επίπεδο τη θάλασσα, θα έχουμε περισσότερη ε, αλλαγή τη στάθμη στην Καραϊβική, αλλά υπάρχουν και ευκαιρίε ευκαιρίες να αλλάξουμε το σύστημα, να έχουμε καθαρότερες θέσει εργασία, να μειώσουμε τη ρήπανση, να έχουμε καλύτερη υγεία και ευημερία και φυσικά να ξεφύγουμε από την ε, ε, εξαιρετική φτώχεια. Όλα αυτά είναι θετικά. Αν γίνουν όλε αυτέ οι αλλαγέ στο αφήγημα, ίσως θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και ε, ο οργανισμός ε, περιβάλλοντος ε, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Η ρήπανση δεν είναι αυτό το οποίο σκοτώνει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να εκριζώσουμε το θάνατο από την πολιομιαλίτιδα, από την ηλαρά ή από την ελονοσία, ε, αλλά η απο την ελονοσια αλλα η ρηπανση δεν είναι ο μεγαλύτερος δολοφόνος ανθρώπων. Πρέπει να μειώσουμε τη ρήμαση όμως για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κλιματική αλλαγή και αντιστρόφως. Αλλά ορισμένες φορές ε, θα πρέπει να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στη ρήπανση. Ε, το αποτέλεσμα είναι άμεσο και ο κόσμος το νιώθει και υπάρχουν και συγκεκριμένες κινήσεις ε, ε και και μπορεί να υπάρξει και μία ε, ραγδαία αύξηση σε κάποιες πόλεις και έτσι να βρεθεί στην πρώτη προτεραιότητα. Η συμβουλή μου είναι να συνεχίσουμε το ίδιο φύγμα που έχουμε στο παρελθόν, αλλά είναι πιο θετικό, να πιστιάζει περισσότερο στην υγεία και να είναι πιο κοντά στους ανθρώπους και να ε, ε, βασιζόμαστε σε συγκεκριμένα στοιχεία. Επίσης, να πω κάποια πράγματα για τους βασικούς στόχους, τους οποίους πρέπει να τονίσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Ο πρώτος είναι η ενέργεια. Χρειαζόμαστε αλλαγή ε, της χρήσης ενέργειας. Έχει αρχίσει, αλλά είναι πολύ βραδία η όλη διαδικασία. Το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά που είχα είχαμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και περισσότερο ηλεκτρισμό από ηλιακή ενέργεια και από τις υπόλοιπε ε, μορφές, αλλά ε, πρέπει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Το 50% αυτών των λαγών δεν μπορούν να γίνουν από μόνες τους. Πρέπει λοιπόν εδώ η Ευρώπη να βοηθήσει και έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα και έχει συμβάλει ουσιαστικά είχαμε ε, τη Γερμανία, για παράδειγμα, πέρσι, που είχε 100% ανανεώσιμες στο ενεργειακό της μείγμα. Και αυτό είναι ε, θετικό, αλλά πρέπει να επιτυχύνουμε. Αν θέλετε θετικά παραδείγματα, το Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα η οποία ήταν κέντρο της βιομηχανικής επανάστασης για ένα και μόνο λόγο, διότι έχει αυθονία άνθρακα, ε, υπήρχε κάρβουνο παντού και φυσικά υπήρχαν και τρόποι να μεταφέρεται το κάρβουνο. Αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μόνο 2% στο ενεργειακό του μείγμα άνθρακα άνθρακα σχεδόν δεν θα χρησιμοποιούν καθόλου και φυσικά ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια συμμαχία κατά τη χρήση άνθρακα και πρέπει να βοηθήσουν και είναι θετικό. Αφού τα κατάφερε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, μπορεί να γίνει σε όλε τι υπόλοιπε χώρε. Το μείγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ηλιακή ενέργεια, υπάρχουν ε, τεράστια αεολικά πάρκα στη Σκοτία, φυσικό αέριο, είναι μείγμα διαφόρων πηγών και όλα αυτά έχουν αντικαταστήσει την πιο ρηπογόνο πηγή. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες ε, επιτυχημένες ε, ιστορίες. Η Δανία, ε, η Κίνα χρησιμοποιεί ηλιακή και ολική ενέργεια και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά και να επιταχύνουμε και τις αλλαγές πολύ γρήγορα. Ένας πολύ σημαντικό τομέα, τον οποίο υποτιμούν οι άνθρωποι, είναι η ψήξη. Πολύ σημαντικό σκέλος της ενέργειας που χρησιμοποιούμε παγκοσμίω είναι για ψήξη. Στη χώρα μου, στην Νορβηγία, έχουμε μία από τις πιο προεδευτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ε, έφτιαξαν ένα πρότυπο κτίριο και μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή στη θερμοκρασία στην Νορβηγία είναι πάνω από τους μείον 5 βαθμούς, που συνήθως είναι, είτε το πιστεύετε είτε όχι, ε, μας ενδιαφέρει η ψήξη και όχι η θέρμανση. Πρέπει να ε, το κτίριο όταν η θερμοκρασία είναι ακόμα και κάτω από το 0 και γιατί αυτό, γιατί όλος ο εξυπλισμός και όλοι οι άνθρωποι παράγουν ενέργεια μέσα στο κτίριο, όλα τα, ε, ε, ε όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής ε, παράγει ενέργεια και επομένως πρέπει να ψύχεται το κτίριο ακόμα και αν έχουμε θερμοκρασία θερμοκρασίες υπό το 0 ε, ε, έξω. Ε, επίσης, Στη Βόρεια Ινδία οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 45 βαθμούς ε, Χρειαζόμαστε λοιπόν συστήματα ψήξη. Ε, Δεκάδε εκατομμύρια άνθρωποι λοιπόν στι επόμενε δεκαετίε θα χρειάζονται περισσότερο ψήξη. Αν γίνουν αυτά με τι παροχημένε τεχνολογίε που είχαμε στο παρελθόν, απαιτούν τεράστια ποσοστά ενέργεια. Κάποιοι προσπαθούν να τα υπολογίσουν όλα αυτά για να δούμε πόσα χρειαζόμαστε για ψήξη και είναι τεράστια τα ποσά. Βεβαίω ε, ε, είναι διαθέσιμη νέα τεχνολογία την οποία μπορούμε να βοηθήσουμε να εξαπλωθεί και να παράγουμε την ίδια ενέργεια με πολύ λιγότερη χρήση ε, ενέργειες και πολύ λιγότερες εκπομπές ε, οι οποίες είναι ρηπογόνες για το κλίμα. Ε, ο Διεθνής Οργανισμός λοιπόν περιβάλλοντος και άλλοι οργανισμοί θα πρέπει να ξεκινήσουν μια μαχία για την ψήξη. Ίσως μπορεί να γνωρίζετε, υπάρχει και το σχετικό πρωτόκολλο για την καταπολέμηση την στρίπα του όζοντος και αυτό έγινε με εξαιρετικό τρόπο και πρέπει να εισαγάγουμε όμως και τις νέες τεχνολογίες ε, που να μην έχουν αρνητικές συνέπειες για το κλίμα για να μπορέσουμε να ε, μειώσουμε και τον αντίκτυπο από αυτά. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε όλες τις αρνητικές συνέπειες για το κλίμα που ε, προκύπτουν από τις, τον εξοπλισμό ψήξης και κατάψυξης που αγοράζεται σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να είναι λοιπόν πιο ενεργητικά αποδοτικά όλα αυτά τα μηχανήματα και αν έχουμε πιο καθαρά συστήματα ψήξη, θα έχουμε και μείωση της υπερθέρμανση. Μειώσαμε την υπερθέρμηση μέσω της αλλαγή του Κιώτα. Μπορούμε να έχουμε άλλο μισό βαθμό μείωση, απλώς παρέχοντα ε, καθαρότερες μορφές ψήξη ε, σε όλο τον κόσμο και φυσικά ε, να μην έχουμε παραδοσιακές μορφές ψήξη στην Ευρώπη. Μπορεί να φαίνεται κάτι μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Η ενέργεια λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε και κυρίως θα πρέπει να δράσουμε και στον πραγματικό κόσμο εκτός ε, και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα μέσω των αποφάσεών μας. Οι Ευρωπαίοι έχουν ε, μεγάλους συμμάχους ανά τον κόσμο. Ο πρόεδρος Μακρόν της Γαλλίας με τον ε, Υπουργό Ίντα είχαμε και προέδρου και αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων από διάφορα μέρη του κόσμου. Εκεί ε, διαμορφώθηκε μια διεθνή συμμαχία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ηλιακή ενέργεια και να είναι στο ενεργειακό μείγμα σε όλο τον κόσμο σε πολύ ε, γρήγορα χρόνους ε, και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνιμη συμμαχία στην Αφρική. Ε, όλοι στην Αφρική όμως έχουν ε, κινητό τηλέφωνο για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται ε, και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη χρήση ηλιακής ενέργειας στην Αφρική ε, διότι αυτή τη στιγμή είναι μικρή η χρήση. Είναι κρίσιμο τομέα λοιπόν η ενέργεια. Ένας άλλος κρίσιμος τομέας, αν δούμε τα στοιχεία, είναι η χρήση γεών και δασών. 20% ε, των εκπομπών του κλίματος ε, είναι από αρνητική χρήση γεών ή από αποψήλωση δασών. Και οι αριθμοί φυσικά είναι πολύ εντυπωσιακοί. Ε, βρήκαμε ε, η τύρφη είναι τεράστια σε ποσότητα, υπάρχουν ε, τεράστια αποθέματα άνθρακα που είναι αποθηκευμένα σε αυτές τις τύρφες ε, και αυτό είναι 20 χρόνια παγκοσμίων εκπομπών από όλες τις πηγές. Εάν λοιπόν αυτά αποδεσμευθούν, για παράδειγμα υπάρχει καύση και χρησιμοποιηθούν στη Γεωργία, θα έχουμε τρία χρόνια παγκοσμίων εκπομπών ή όλες οι εκπομπές των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος βεβαίως ότι αυτές οι περιοχές θα καούν, αλλά ε, ε, με τις εξελίξεις που έχουμε ε, στο Κονγκό ε, και στις δύο χώρες του Κονγκό θα ε, μπορέσουμε να, μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα. Είναι σε ένα πολύ απομακρυσμένο τμήμα, πολύ κατοικημένο αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να αρχίσει προστασία σε έγκαιρο, εγκαίρος για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πράγματα. Έχουμε και μια συμμαχία με την Ινδονησία που είναι η χώρα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε θέματα τύρφης και οι δύο χώρες του Κονγκό και η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα μπορούσε να συμμετέχει και ως εταίρος όλα αυτά. Οι πολιτικές λοιπόν βοηθούν στον τομέα αυτό. Η Βραζιλία έχει μειώσει το ποσοστό της αποψήλωσης του Αμαζονίου κατά 40%. Ε, κάποιοι μπορεί να πούνε ότι πρέπει να αυξηθεί και άλλο αυτό, αλλά ε, υπάρχει μεγάλη μείωση στην αποψήλωση. Ε, αλλά υπάρχει και ε, κάποια αύξηση σε κάποια σημεία. Δεν είναι απόλυτα γραμμική η διαδικασία. Ε, εκεί που μειωνόταν, ξαφνικά η αποψήλωση αυξήθηκε στον Αμαζόνιο, στη Βραζιλία και μετά ξαναέπεσε. Πιστεύω ότι είναι αξιοσημείωτο το αποτέλεσμα. Είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται σε πλήρη πολιτική παράλυση. Υπάρχει απόλυτη κρίση. Κανεί δεν ήξερε ποιο ε, θα είναι ε, πρόεδρο τον Οκτώβριο. Δεν γνωρίζει κανεί ακόμα. Και είναι και όσο το δυνατόν πιο σκληρή η πολιτική μάχη στη χώρα. Και μόνο το γεγονός όμως ότι είτε η αριστερά είτε η δεξιά κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση για τον αποψήλωση του Αμαζονίου είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ε, σημάδι ότι έχει πλέον περάσει στο DNA των Βραζιλιάνων αυτό. Στο μέλλον η Βραζιλία που είναι η μεγαλύτερη ε, δασική χώρα έχει δείξει στις υπόλοιπες χώρες τι μπορεί να κάνει. Να περάσω τώρα στην Ινδονησία ως παράδειγμα. Σε ό,τι αφορά την έγκριση όλων των νόμων ε, που επιθυμούμε και ε, παρά τις δραστές έγκριπες ε, Βέβαια, οι από τους νέους νόμους πέρασαν και από το Κοινοβούλιο και έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό και από την κυβέρνηση και στην Ινδονησία και στη Σιγκαπούρη όλες οι σχετικές επιχειρήσεις υλοτομίας έχουν, προσπαθούν να συμβάλλουν ε, στην ε, καταπολέμηση τη αποψήλωση. Οπότε λοιπόν παρότι υπάρχει ε, συμφωνία και σε πολιτικό επίπεδο και βούληση σε οικονομικό επίπεδο, δεν επιτυχάνουμε μείωση τη αποψήλωση γιατί υπάρχουν πολύ χαμηλά κίνητρα σε τοπικό επίπεδο να γίνουν σεβαστοί αυτοί οι νόμοι της αποψήλωσης. Δηλαδή υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Ε, πώς θα καταφέρει να επανεκλεγεί. Μπορεί να επιτρέψει κάποιο είδους τέτοιους, τέτοιους δράσεις. Δίνει τέτοιου είδους άδειες για παράδειγμα. Δηλαδή Ε, και αν ε, μπορεί κανείς να αποψηλώσει το δόση ώστε να δημιουργήσει περισσότερους, ε, περισσότερα εδάφια κατοικήσιμα μπορεί να επανεκλεγεί. Άρα λοιπόν ποια θα πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση θα πρέπει να καλέσουμε τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν την νομοθεσία αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μετασχηματίσουμε δυνατή τις τοπικές οικονομίες έτσι ώστε οι άνθρωποι εκεί οι κάτοικοι να επωφεληθούν από τη μείωση της αποψήλωσης. Αν δουν δηλαδή οι άνθρωποι ότι τελικά η καθημερινή του ζωή βελτιώνεται με τη διατήρηση των δασών ε, θα συμβάλλουν σε αυτό. Όλη η εμπειρία μας μας δείχνει ότι όταν οι άνθρωποι υπερασπίζονται ε, το, το, το δικό τους χώρο, το δικό τους δάσος σε τοπικό επίπεδο, έχουμε την καλύτερη δυνατή εγγύηση για την προστασία αυτού του δάσους. Ε, στη Βραζιλία αυτή η πολιτική ήταν πολύ ε, σημαντική. Δηλαδή αυτή η, αυτό το μήνυμα που πέρασε στους Ιθαγενείς ε, εκεί προκειμένου να περασπιστούν τα δάση τους. Ε, στην Ινδονησία λοιπόν έχουμε ξεκινήσει, ε, έχει ξεκινήσει με την BNP Παριμπά και άλλους πολύ σημαντικούς εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή προσπάθεια, μια συσπήρωση δυνάμεων έτσι ώστε να επενδύσουμε στην βιώσιμη γεωργία και στην Ινδονησία αλλά και στην Ινδία έτσι ώστε για παράδειγμα οι καλλιεργητές ε, φοινικότητων ε, να μπορέσουν να βελτιώσουν την ε, παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους έτσι ώστε να μην θέλουν να προβούν σε περισσότερη αποψήλυση των δασών. Άρα λοιπόν υπάρχει περισσότερο δυναμικό να, να, να, δοθεί, να, να επιτραπεί περισσότερη παραγωγικότητα αντί να καταστρέφονται τα δάση. Και από εκεί και μετά θέλουμε μια, ένα τέτοιο συνδυασμό. Δηλαδή από τη μία πλευρά εφαρμογή της νομοθεσία σε κρατικό επίπεδο και παροχή κινήτρων σε τοπικό οικονομικό επίπεδο. Ένα τέτοιο συνδυασμό είναι πολύ επιτυχημένο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράσχει και οικονομική υποστήριξη. Το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά κάποια χρηματοδότηση θα μπορούσε να δώσει την όθηση για να λάβει χώρα αυτή η αλλαγή. Ε, και να σα πω ε, κάτι, ότι μία σημαντική οικονομική πηγή ε, για να επιτευχθεί αυτό είναι ε, η εφαρμογή του συστήματος εμπορία εκπομπών από το 2020 στην αεροπορία. Κάτι τέτοιο είναι πραγματικά φανταστικό γιατί εάν υπάρχει μία ε, βιομηχανία η οποία μοιραία θα αυξήσει τις εκπομπές της είναι η αεροπορία. Ε, και 50 εκατομμύρια από το τρία συνολικά δις που έχουν προκύψει σε αυτό το τομέα προέρχονται ακριβώς από το τομέα της αεροπορίας. Και η Κίνα αναφέρει ότι 400 ε, εκατομμύρια έχουν μπει στα από αυτό το σύστημα, οπότε ε, βλέπουμε ε, πολύ μεγάλη αύξηση της αέριας κυκλοφορίας και κατά συνέπεια αναμένουμε πολύ υψηλά έσοδα για το σύστημα εμπορίας εκπομπών και θέλουμε ένα τμήμα αυτών των κοντιλίων να, να κατευθυνθεί προς την προστασία των δασών. Δηλαδή, ε, ένα περιοδικό που έχει κανεί, ε, για παράδειγμα στα αεροσκάφη μπορεί να το γεμίσει ακριβώς ε, με φωτογραφίες από κορίλε ή από τα παρθένα για παράδειγμα δάση της Βραζιλία. Οπότε θα γίνουν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα χρειαζόμαστε να ε, δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις που θα γίνονται από τα έσοδα του συστήματος εμπορίας να γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και να ε, οδηγούν σε αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα συντομία σε δύο ακόμα ζητήματα. Τα πλαστικά έχουν αναφερθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα εδώ και έχει γίνει φανταστική πρόοδο, ειδικότερα το βήμα που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. δηλαδή την ίδια εβδομάδα αποφασίστηκε ε, και η ε, κατάργηση ε, των πλαστικών στο 2022, πράγμα το οποίο βέβαια Ε, πολύ δύσκολο να βγει κανεί, ε, για παράδειγμα, στο Βρετανικό ή Γαλλικό Κοινοβούλιο και να πει εμεί ω άλλη χώρα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια κατάρριξη πλαστικών. Κανεί δεν μπορεί να κρυφτεί από αυτή την υποχρέωση. Είναι πραγματικά θετικό το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η παράλληλη ε, πρόοδο και αυτό βέβαια σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή, γιατί η η οικονομία η οποία ε, θα αξιοποιήσει και θα ανακυκλώσει αυτό το πλαστικό είναι και πολύ πιο ε, φιλική προ το περιβάλλον. Όλο αυτό το πλαστικό που θα ανακυκλωθεί θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Ε, Υπάρχει πολύ πλαστικό που χρησιμοποιούμε και δεν το χρειαζόμαστε. Αυτά τα πλαστικά μπουκάλια που βλέπω εδώ μπροστά μου δεν τα χρειάζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να γεμίζετε τα δικά σα μπουκάλια. Ναι, Πρόεδρος λέει ότι ήδη το έχουμε εφαρμόσει, απλά μα έχουν μείνει αυτά τα μπουκάλια ίσως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, κάποιο είδους ε, ATMs, αν θέλετε, μηχανές εντό εισαγωγικών, οι οποίες αντί για χρήματα μας δίνουν νερό. Δηλαδή μπορούν να υπάρξουν τέτοια μηχανήματα, μπορεί να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Και ε, τα πλαστικά λοιπόν αποτελούν ε, τμήμα τη προσπάθεια που θέλουμε κατά την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Τέλο, πρέπει να, να, να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Το 2020 θα λάβει η χώρα η διάσκεψη του Πεκίνου με τα συμβαλόμενα μέρη σε ό,τι αφορά τη βιοπικιλότητα ε, και θέλουμε αυτό να αποτελέσει ένα ερώσιμα για την προστασία τη βιοπικιλότητα και για την προστασία τη άγρια φύση, όπω ήταν ορόσημο για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι. Και υπήρξε και μια συνάντηση με ε, ε, και η, η, στη διάσκεψη του Πεκίνου ε, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία ε, για να ε, γίνει μια αλλαγή της πολιτικής στην Κίνα για την οποία θα χρειαστεί την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η πολιτική δηλαδή βούληση που είναι απαραίτητη εδώ προέρχεται από τη Ουάσιγκτον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βρυξέλλες και τα άλλα κράτη-μέλη και από το Πεκίνο, από την Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος ε, για αυτή την ενημέρωση από τον κύριο Ζόλκαμς ε, ως προς τα όσα συμβαίνουν ανά τον κόσμο σε σχέση με αυτέ τι πολιτικέ. Και τώρα, συνάδελφοι, ποιοι θέλετε να πάρετε το λόγο, ο κύριο Λάινεν. Ο κύριος Λάινεν λοιπόν πρώτο, παρακαλώ. Ναι, Έρικ, ε, σε ξέρω εδώ και καιρό. Ελτήρια για τον αραβόνα σου και για τις δεσμεύσει σου, ε, για την ε, αφοσίωσή σου. Ε, δεν βλέπουμε τόσους πολλούς ηγέτες τόσο συχνά που δεσμεύονται τόσο έντονα και τους ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό που κάνουν. Ε, το ΟΗΕ ε, στο δικό σου τον κλάδο εξελίχθηκε από πρόγραμμα σε πραγματική, αυθεντική και αυτόνομη οργάνωση. Ε, είναι ενδιαφέρον γιατί θα βοηθήσει κυριολεκτικά την, τον πλανήτη. Ε, ένας από τους στόχους είναι ένας πλανήτης χωρίς μόλυση. Ε, για να προωθήσουμε τον, τον αγώνα κατά της ε, κλιματικής αλλαγής χρειαζόμαστε ένα αφήγημα το οποίο να είναι προσιτό, να το καταλαβαίνει κάθε πολίτης σε κάθε χωριό, σε κάθε περιοχή, σε κάθε πόλη. Φυσικά είμαστε αργοί. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε το ψήφισμά μας για το Κατόβιτσε και πάλι παραπονιόμασταν ότι είμαστε αργοί. Υπάρχουν οι τεχνολογίες. Συχνά η χρηματοδότηση των ε, αλλαγών και των μετασχηματισμών λείπει πράσινη χρηματοδότηση. Υπάρχουν τόσα πολλά λεφτά στον κόσμο. Πώς θα βρούμε περισσότερα λεφτά για πράσινους σκοπούς. Δεύτερο ερώτημα αφορά την προσαρμογή. Μένω κοντά στο Λουξεμβούργο. Και εκεί είχαμε τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες ε, τρεις φορές ε, κυκλώνες. Πρέπει να προσαρμοστούμε και η UNEP. Πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Ε, δηλαδή το θέμα της προσαρμογής στα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσου. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Οπότε, το πρώτο μου ερώτημα είναι το εξής. Σε ό,τι αφορά την ε, Συμφωνία των Παρισιών, υπάρχουν εδώ συγκεκριμένες ε, νομικά δεσμευτικές ε, συμφωνίες στις οποίες έχουμε καταλήξει, δεσμεύσεις δηλαδή από την πλευρά των 100 μελών, αλλά ο κ. Σιμπράντη είπε και προηγουμένως ότι τελικά δείχνουν να μην είναι δεσμευτικές αυτές τις συνεισφορές. Και ε, ειδικότερα σε σχέση με αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα καταφέρουμε να θέσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε ενώπιον των εθνών τους. Δηλαδή ο πρόεδρος Ομπάμα είχε αποδεχτεί συγκεκριμένε ευθύνε για την αμερικανική πλευρά, ε, τις οποίες τώρα δεν θέλει να εφαρμόσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αξιώσουμε από την Αμερική να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Δεύτερο ερώτημα. Ε, σε ό,τι αφορά τον στόχο των δύο ε, βαθμών Κελσίου, να πω ότι ε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το 10% των εκπομπών. Αν κάνουμε λοιπόν εμείς από την πλευρά της Ένωσης ό,τι χρειάζεται για να επιτύχουμε έστω και τον 1,5 βαθμό, παρόλα αυτά δεν θα συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα από την πλευρά των κρατών τα οποία δηλαδή ε, ε, είναι υποχρεωμένα να εξετάσουν και περαιτέρω πτυχέ από την επίτευξη αυτών των στόχων. Ε, με δύο λοιπόν βαθμούς Κελσίου στόχο για τα κράτη-μέλη νομίζω πω είμαστε εντάξει απέναντι στι υποχρεώσει μα, γιατί υπάρχει και οικονομικό και κοινωνικό κόστο για όλα αυτά. Και κάτι ακόμα. Αυτό που είπε και ο επικεφαλή εδώ του προγράμματο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε και θετικοί στι αναφορέ που κάνουμε για το κλίμα. Δεν θα πρέπει δηλαδή πάντοτε να περιγράφουμε εδώ σενάρια τρόμου. Θα πρέπει να είναι θετική, αισιόδοξη προσέγγιση μας. Αυτό παρότι βέβαια ισχύει από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αυταπατώμαστε. Ε, δηλαδή, ε, αν δείξουμε για παράδειγμα ε, το πόσο καταπληκτικά είναι τα όσα συμβαίνουν με αυτό το νέο αεροδρόμιο στην Νότια Ινδία ή το πόσο καταπληκτικά δουλεύουν και συνεισφέρουν στην παροχή ενέργειας στα αεολικά πάρκα, ναι μεν παρουσιάζουμε κάτι καλό, αλλά είναι και κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αέρα πολύ, ας το πούμε έτσι, για ολικά πάρκα έχουμε στην Βόρειο Ευρώπη. Πολύ ήλιο έχουμε στην Νότια Ινδία. Αυτό δεν ισχύει για όλε τι περιοχέ του κόσμου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ σε σχέση με τα όσα ε, παρουσιάζουμε. Εγώ βέβαια πιστεύω πάρα πολύ σαν ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αλλά ε, αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι αιωλικά πάρκα, νομίζω. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Madam Chair. And... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σολχάιν, που ήρθατε εδώ, λέει ο Μπράντι. Είναι σημαντικό να ακούσουμε μια παρουσίαση από εσά που έχετε την εποπτική εικόνα του πράγματος και μας παρουσιάσατε όλα όσα κάνατε. Ε, εστιάστε πολύ στην κλιματική αλλαγή, δικαίω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι τελικά θα βρούμε τεχνολογικές λύσεις για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Και τα παραδείγματα του Μουσείου Άνθρακα του Κεντάκη είναι εντυπωσιακό. Ε, συμφωνώ μαζί σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Αναφέρατε τον Τραμπ. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ δεν είναι ο λόγος του προβλήματος στις ΗΠΑ. Είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης προσπάθειας και κινήματος ανθρώπων και στην Ευρώπη υπάρχει αυτό και σε άλλα μέρη του κόσμου που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι πιστεύουν πραγματικά ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Απλώς θοκαμιλίζουν και προσπαθούν να αποφύγουν να το σκεφτούν αυτό το πρόβλημα. Ψάχνουν να βρουν πολιτικές λύσεις που είναι εντελώς βαχυπρόθεσμες και που τελικά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό γιατί νομίζω ότι είναι μείζον. Μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η δημοκρατία που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να αντιμετωπίσουμε τέτοια μεγάλα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια διοπικιλότητας και άλλου τέτοιου τύπου προβλήματα. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε δημοκρατία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά πώς θα το κάνουμε ούτω ώστε να πιστέψει η πλειοψηφία του, των ανθρώπων στην, στην ατζέντα μας. Ε, δεύτερον, αναφερθήκατε στη βιοπικιλότητα, την απόλυτη την αποψήλωση των δασών. Είναι μια σιωπηλή κρίση. Όλοι μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, αλλά μιας να ξεχνάμε τα τεράστια προβλήματα απώλειας της βιοπικιλότητας που έχουν από πίσω. Φοβάμαι ότι η ανθρωπότητα θα πεθάνει πριν από την κλιματική αλλαγή λόγω της α, α, έλλειψης βιοπικιλότητας. Τόσο επίγον το θέμα. Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρω το CBD δουλεύει, ασχολείται με αυτό. Και η κόπα του 2020 στην Κίνα θα είναι πολύ σημαντική για αυτό το πράγμα. Ε, το βασικό πρόβλημα είναι η αύξηση του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που όλοι το βλέπουμε και κανένα δεν το λέει. Δείτε στην Ασία, αλλά κυρίω στην Αφρική σε ευαίσθητες περιοχές. Ε, αναμένουμε αύξηση του πληθυσμού. Είναι σαν να ε, προσπαθούμε να κερδίσουμε μια μάχη όπου αλλάζουν οι στόχοι. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε για την κλιμαλλαγή, αλλαγή, αλλά πιστεύω και πιστεύω ότι θα βρούμε τεχνολογικέ λύσει γι' αυτό, αλλά τι θα γίνει με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Απόλυτη επικοινότητα, αποψήλωση των δασών κτλ. Αν δείτε επίση την τεράστια αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού σε χώρε όπω η Νιγηρία και σε άλλα μέρη τη Αφρική. Χρειαζόμαστε πολιτικέ για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αύξηση του πληθυσμού και να βρούμε λύσει δεδομένη αυτή. Όχι, πρέπει να σταματήσει αυτή η αύξηση του πληθυσμού τι επόμενε δεκαετίε. Είναι πολιτικό ταμπού, το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το δεύτερο ερώτημά μου. Με ποιο τρόπο η οργάνωσή σα, στο UNEP μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Ζολχάιμα για αυτήν την ε, καταπληκτική παρουσίαση που μας κάνατε. Θα ήθελα να θέσω δύο-τρία ερωτήματα. Σε γενικές γραμμές η εντύπωση που είχα από την, παρουσίασή σας, από την παρουσίασή σας ε, είναι ότι έχουμε μια γενική εικόνα, για μια γενικά καλή εικόνα σε ό,τι αφορά ε, τα αρχικά βήματα που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά έχουν έτσι τα πράγματα, γιατί κάθε χρόνο ακούμε να επιτυχάνουμε ένα υψηλότερο κάθε φορά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τις εκπομπές άνθρακα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο τώρα ερώτημα. Αναφερθήκατε κυρίως στην ενέργεια, αλλά και στη χρήση των εδαφών, πιο προσεκτικά βέβαια, αλλά δεν αναφερθήκατε συγκεκριμένα στην γεωργία. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθούν ε, στην ε, ε, έκθεση του κύκρου του κύριου Χένινγκ από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά την γεωργία. Εδώ λοιπόν έχουμε μία δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια μας γιατί βλέπουμε ότι έχει παρατηρηθεί μέσα το 2005 μια, ένας διπλασιασμός της παραγωγής κρέατος και η έκθεση του δόκτωρου Στάινφελντ είχε τότε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 18,2 των εκπομπών ε, σήμερα στον κόσμο προέρχεται από το τομέα της γεωργίας και συγκεκριμένα από το κλάδο της παραγωγής σε κρέατος. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Κίνα προέβησε κάποια σημαντικά βήματα κατά την τελευταία διάσκεψη κορυφής. Η Κίνα ανέφερε ότι θα ήθελε να μειώσει την κατακεφαλή κατανάλωση κρέατος Ε, σε 45-75 γραμμάρια ε, ε, την ημέρα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία αντίδραση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, άλλε περιοχέ του πλανήτη δεν αντιδρούν σε μια τέτοια βούληση τη Κίνα. Άρα, λοιπόν, το πρόβλημα τη παραγωγή κρέατο δεν αναφέρθηκε από τη δική σα πλευρά, κύριε Ζόλχαμ, και θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση Και από εκεί και μετά σε ό,τι αφορά την αποψήλωση των δασών και την ε, μείωση της βιοπικιλότητας. Εγώ συμμετέχω στις ε, εργασίες της ε, Επιτροπής για την Νοτιοανατολική Ασία και δεν διαπιστώνω ότι η βούληση των κρατών αυτών είναι να σταματήσουν την αποψήλωση των δασών. Ο στόχος του είναι απλά να μειώσουν τους ρυθμούς της αποψήλωσης των δασών. Το ίδιο συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή έχουν μειωθεί οι ρυθμοί της αποψήλωσης των δασών αλλά δεν έχουν σταματήσει. Πώ θα καταφέρουμε λοιπόν το να σταματήσει, να τερματιστεί η αποψήλωση των δασών. Γιατί νομίζω πω αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχο. Πλήρη ε, διακοπή τη ε, μείωση των δασών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο σε εσά, κύριε Σόλχαϊμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω μία προς μία. Ε, και εγώ θα προτιμούσα, κύριε Λάινεν, να είναι οργανισμός ε, η υπηρεσία, αλλά δεν θα χάσω χρόνο. Γι' αυτό σημασία έχει να τα καταφέρουμε για το κλίμα και το να δίνουμε μάχες οι οποίες ε, θα είναι καταδικασμένες στην αποτυχία δεν θα οδηγήσει και τίποτα. Ε, ο η διαφορά μεταξύ οργανισμού και προγράμματος δεν είναι μεγάλη. Εγώ ούτως ή άλλως αφιερώνω το χρόνο μου ε, να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά για να το καταλάβει ο κόσμος ε, τι συμβαίνει για το περιβάλλον και όλοι το καταλαβαίνουν όταν αναφέρομαι στα ε, πρόγραμμα των ΕΕ για το περιβάλλον. Αν μπορέσετε να το διορθώσετε, Πείτε μας πώς θα το διορθώσουμε, αλλά να μην εστιάζουμε στα εσωτερικά θέματα των Εθνών, αλλά στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη, την Αφρική, την Κίνα και τους υπολείπους να έχουν ένα ε, πλανήτη χωρίς ρήπανση μας ενδιαφέρει η χρηματοδότηση και πρέπει να έχουμε ε, δυνατότητα να κινούνται τα χρήματα να τον κόσμο προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πολύ εστιαστεί στην ανάπτυξη και στη συνδρομή και ξέρετε ότι υπάρχει θέμα ανακτηξιακής βοήθειας, αλλά είναι ελάχιστα τα ποσοστά. Ακόμα και στην υποσαχάρη Αφρική οι επενδύσεις είναι κάτω από το 5% της οικονομίας. Η ανάπτυξη δεν έχει διαδραματίσει κανένα ρόλο στην ε, εξέλιξη της Κίνας. Επομένως, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 100 φορές πλουσιότεροι στην Κίνα από τους γονείς τους, ούτε καν τους παππούδες τους, από τους γονείς τους από τότε που ξεκίνησε η εξέλιξη της Κίνας. Το θέμα είναι λοιπόν να έχουμε τη σωστή πολιτική, να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα και όχι ε, να αναπτύξουμε την, ε, ε, την αναπτυξιακή βοήθεια. Μπορεί να αποτελέσει καταλήτη σε κάποιες περιοχές, αλλά δεν βοηθά και απαραίτητα. Επίσης, πρέπει να καθορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε βοηθήσει και ασφαλιστικές εταιρείες. Τώρα έχουμε τις μεγαλύτερες τράπεζες ανά τον κόσμο. Κάποιες τράπεζες έχουν προσυπογράψει. Έχουμε τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Κίνας η οποία θα συμμετέχει και ε, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. και να περάσουμε πραγματικά στην πράσινη οικονομία. Και φυσικά το πρόγραμμά μας ήταν πολύ σημαντικό και είναι κεντρικό και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν ε, και μεγάλες τράπεζες, ε, η Χαμπρομπάκ των κάτω χωρών που έχουν ε, συστήσει ιδιωτικά προγράμματα για ιδιωτικές επενδύσεις και δούμε, να δούμε πώς μπορούμε να αντιλήσουμε και διδάγματα και να τα αντιγράψουμε όλα αυτά και σε άλλες περιπτώσεις. Κύριε δεν μπορούμε να στείλουμε την αστυνομία να ε, παρακολουθεί τι Ηνωμένε πολιτείε και να τι υποχρεώσει να τηρούν ε, διεθνεί ε, υποχρεώσει ούτε την Πολωνία. Το θέμα είναι πολιτική εξουσία και η σωστή πολιτική για το κλίμα σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές, όλη η πολιτική και όλα τα κράτη καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό και δεν το κάνουν για κάποιον άλλον, το κάνουν για τη δική του τη χώρα. οι νομικά δεσμευτικέ συμφωνίε βέβαια πάντα είναι η προτιμητέα λύση, αλλά ορισμένε φορέ και οι μη δεσμευτικέ λύσει μπορεί να αρκούν αρκεί να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή. Αναφερθήκατε στη Γερμανία. Εγώ όταν ταξιδεύω ανά τον κόσμο πάντα αναφέρομαι στη Γερμανία. Το έκανα και την περασμένη εβδομάδα και τη δίνω ως παράδειγμα. Διότι κάποιοι λένε ότι υπάρχει αντάλλαγμα μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και σοβαρής εμπλοκής με το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται μακρά απάντηση. Μπορείς να πεις όχι. Ορίστε η Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι ίσως η χώρα στον πλανήτη που έχει κάνει εσκεμμένες αποφάσεις για πράσινη οικονομία. Ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, ένα περιοδικό ε, κατέταξε όλες τις χώρες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές και οικονομικές τους επιδόσεις και είπαν ότι η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση. Και επειδή αναφερθήκατε και στην Νορβηγία, να σας πω ότι μπορεί η κατάσταση σε, να είναι καλύτερα από την Νορβηγία, αλλά είναι τυχερή, είναι λιγότεροι Νορβηγοί. Έχουμε 80 εκατομμύρια Γερμανούς και 5 εκατομμύρια Νορβηγούς. Ε, οι Γερμανοί συνειδητά έχουν λάβει αποφάσεις ε, να περάσουν προς ε, μια πιο οικολογική οικονομία, χάρη στην κοινωνία, χάρη στο γεγονός ότι και η Άγγελα Μέρκελ και ο υπερβολικός υπουργό Περιβάλλοντος, που είναι πολύ σημαντικός για αυτήν, και οι σοσιαλδημοκράτες ήταν ε, υπέρ των ε, πολιτικών αυτών και επίση οι πολίτες και το κόμμα των Πρασίνων πρόθεσαν τα θέματα αυτά. Και ε, αυτό είχε καλύτερα αποτελέσματα για τους Γερμανούς, όχι μόνο για την φύση, αλλά και για τις θέσεις εργασίας. Και η κυρία Μέρκελ πηγαίνει ανά τον κόσμο και προωθεί πολλές επιχειρήσει που σχετίζονται με ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και περιβαλλοντική προστασία, γιατί ε, ορισμένες φορές τα αιτήματα ήρθαν από την κοινωνία των πολιτών. Μετά πέρασε στη γερμανική κοινωνία γενικότερα και οδήγησε και σε θέσει εργασία και σε οικογένειακέ επιχειρήσει σε όλη τη Γερμανία. Είναι παράδειγμα λοιπόν η Γερμανία είναι απάντηση γι' αυτό, αλλά σύντομα και η Κίνα θα είναι απάντηση. Δεν υπάρχει λόγος να ανταλλάξουμε την ανάπτυξη με το περιβάλλον, μπορούμε να καταφέρουμε και τα δύο. Τώρα, κατά πόσο η δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον θέμα. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία είναι το πιο ε, ηθικά ανώτερο σύστημα ανά τον κόσμο. Αν ρωτήσει τον κόσμο ποιο είναι το καλύτερο σύστημα, οι περισσότεροι θα σου απαντήσουν η δημοκρατία. Αλλά το θέμα είναι αν μπορεί η δημοκρατία να οδηγήσει σε αποτελέσματα. Αν τελικά δηλαδή τα συστήματα, υπάρχουν άλλα συστήματα τα οποία δίνουν καλύτερα αποτελέσματα στον κόσμο, τότε εμεί θα έχουμε αποτύχει ω Ευρωπαίοι. Διότι αν ρωτήσουμε ποιο είναι καλύτερο καλύτερο σύστημα. Ε, θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να δίνει αποτελέσματα στην εκπαίδευση, στην υγεία, στο περιβάλλον, σε καλύτερη ζωή. Και επομένω η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει και πρέπει να απαντήσει καταφατικά. Ναι, η δημοκρατία μπορεί να ε, δώσει αποτελέσματα γιατί τελειώ θα είναι τεράστια αποτυχία. Ο λόγο για τον οποίο είναι απελπισμένο ο κόσμο είναι αρνητική εικόνα για τον κόσμο που εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωση. Ε, θα μπορούσα να σα συστήνω βιβλία, αλλά θα μπορούσα να συστήσω ε, να δείτε τον Στίβεν Πίνκερ, τον Αμερικάνο διανοητή, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο διαφετισμός αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει στο βιβλίο του από περίοδο σε περίοδο και δείχνει πώς είναι καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι το παρελθόν ήταν λαμπρές στιγμές και δεν ξεχνάνε, δεν θυμούνται ότι ιστορικά το προσδόκιμο ζωής ήταν 10 ε, χρόνια λιγότερο μέχρι να αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα ε, στο Μάντσεστερ και ε, στα 1870 όλοι είχαν προσδόκιμο ζωής κάτω από τα 40 και ο μέσος όρος παγκοσμίω ήταν τα 29. Τώρα το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι τα 71 χρόνια και οι γυναίκες στην Νότια Κορέα μπορεί να φτάσουν και τα 90. Όχι μία, γιατί αυτό συνέβαινε και παλιά, αλλά κατά μέσο όρο. Επομένως είναι εξαιρετική αυτή η πρόοδος και ο κόσμος ε, δεν το γνωρίζει, τους το κρύβουμε, είναι ένα πολύ καλά κρυμμένο μυστικό. Βέβαια αν πάει κανείς στην Κίνα δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αρνητισμός, αυτό είναι ευρωπαϊκό και αμερικανικό φαινόμενο. Ο κόσμος πιστεύει ότι ο κόσμος γίνεται χειρότερος, ενώ αν πάτε στην Κίνα και στην Ινδονησία υπάρχει ακριβώς αντίθετη στάση, πιστεύουν ότι υπάρχει τεράστια πρόοδος. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την αρνητική νοοτροπία και να επικεντρωθούμε στα θετικά. Και στο περιβάλλον έχουμε πολλά θετικά. Ε, η όξινη βροχή, για παράδειγμα, ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη πριν από 20-30 χρόνια. Έχει εξαφανιστεί. Στη χώρα μου, στην Ορβηγία, η κατάσταση στη φύση είναι η καλύτερη που είχαμε πριν από την, ακόμα και πριν από τη βιομηχανική επανάσταση. Για 100 χρόνια δεν είχαμε ε, σολομό στους ε, ποταμούς μας ε, και από τη ρήπαση από του ποτανούς και από τη ρήπαση που είχαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλε χώρε. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί δραστικά η ρήπαση και οι σολομοί έχουν επιστρέψει σε όλη την νότια Νορβηγία. Είστε πρόσδεξοι να έρθετε να ψαρέψετε το σολομό, έχουμε άφθονο. Και φυσικά ε, υπάρχει το ίδιο και ε, με την υπόγλωσσα. Και άλλη μια επιτυχημένη ιστορία. Και φυσικά ε, θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να ακολουθήσετε την άποψή μου στους δύο ε, περιοχές του κόσμου όπου υπάρχει σοβαρό θέμα για την ανάπτυξη του πληθυσμού. Το ένα είναι η Νότια Αφρική και στις άλλες είναι η Νότια Σφία. Σε όλες τις άλλες περιοχές δεν έχουμε τεράστια αύξηση του πληθυσμού, ίσα ίσα έχουμε μείωση του πληθυσμού. Η Κίνα έφτασε στο Ζενίθ και τώρα θα αρχίσει να πέφτει. Η Ιαπωνία μειώνεται δραστικά, οι Ηνωμένε Πολιτείε μειώνονται δραστικά, επομένως το πρόβλημα είναι κυρίως για την Αφρική και για την Νότια Ασία είναι ιδιαίτερα ε, σοβαρό στην περιοχή του Σαχέλ που έχουμε 7 με 8 παιδιά κατά μέσο όρο σε κάθε γυναίκα και 3 με 4% αύξηση του πληθυσμού. Είναι μία από τις πιο ευάλωτε περιοχές του κόσμου και μία από τι περιοχές που μπορεί να ε, δημιουργήσουν φυσικά και μετανάστες που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Πρόκειται για μία από τι πιο ευάλωτε περιοχέ από πλευρά περιβάλλοντο, ελάχιστε δυνατότητε ε, εργασία, ελάχιστη εκπαίδευση και φυσικά ε, υπάρχει πρόβλημα για τη διαβίωση αυτών των παιδιών και αυτό δεν είναι βιώσιμο από τι άλλε περιοχέ του κόσμου βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αρχίσουν οι γυναίκε να μορφώνονται, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη ε, και μειώνεται δραστικά η αύξηση του πληθυσμού. Στο Ιράν τώρα έχουμε λιγότερο από δύο παιδιά ανά γυναίκα. Ε, στο Μπαχρέιν είμαστε στο 2,3-2,4 που είναι το σωστό ποσοστό αύξηση πληθυσμού. Εξαιρετική πρόοδο και θα θυμάστε ε, ότι το Μπαγκλαντές ήταν ε, ε, αποτυχημένη περίπτωση. Τώρα είναι μια χώρα που έχει προβλήματα, αλλά έχει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερο κοινωνικό σύστημα και φυσικά η αύξηση του πληθυσμού είναι απόλυτα σταθερή. Βελτιώνεται έτσι η κατάσταση των γυναικών όταν εκπαιδευτούν. τότε υπάρχει οικονομική αύξηση. με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τον πληθυσμό. Και στην Αφρική ο πληθυσμός ε, είναι σταθερός. Σε κάποια μέρη όμως Αφρικής ε, είναι τεράστιο θέμα και η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προστατευτεί μόνο με φράχτες. Θα πρέπει να δει πώς θα βελτιώσει ε, τις ε, συνθήκες διαβίωσης και στην Ευρώπη και εκτός. Ας πούμε στο Σαχέλ μπορούμε να αξιοποιήσουμε την περιοχή εκεί για ηλιακή ενέργεια. Έχει συνέχεια ήλιο. Ε, όταν με αυτόν τον τρόπο, όταν χρησιμοποιούμε το, την ενέργεια αυτή, μπορούμε να αντλήσουμε νερό για να κάνουμε πιο πράσινη την περιοχή. Φυσικά δεν μπορούμε να τα αντιγράψουμε αυτά πάντα παντού, ε, από το ένα μέρο στο άλλο. Ε, γεωργία, τεράστιο θέμα για το κλίμα και το περιβάλλον, για τη βιοπικιλότητα και πολύ από την απώλεια της βιοπικιλότητας οφείλεται στις μονοκαλλιέργειες. Ε, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μέλισσες, που ήταν πολύ θετική πρωτοβουλία. Ε, χρειαζόμαστε και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες και πρέπει να περάσουμε σε ένα είδος γεωργίας που να είναι να βασίζεται λιγότερο στις μονοκαλλιέργειες. Κάτι άλλο, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία στο Ίντρα στην Νότιο Ινδία, είναι βασίζω, ε, μετασχηματίζουμε τις μονοκαλλιέργειες σε ε, καλλιέργειες που είναι πιο φυσικές, ας πούμε, 150 ε, εκμεταλλεύσεις ε, που είναι τεράστιες εκτάσεις αυτές. Ε, είναι όλες οι γεωργικές εκτάσεις ας πούμε της Σκανδιναβίας μαζί. Εκεί λοιπόν αποφεύγουμε και τα χημικά και τα λιπάσματα. Η αποφορά που είχαν αυτά τα εδάφια ας πούμε έχει μειωθεί πάρα πολύ και λιγότερα βεβαίως, πολύ λιγότερα φυτοφάρμακα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και το ξέρω ότι η γεωργία είναι τεράστιο θέμα για το μέλλον. Θα χρειαστούμε πολύ περισσότερα τρόφιμα. Ο πληθυσμός ε, τα επόμενα χρόνια θα φτάσει στα 9,5 δισεκατομμύρια με 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για 2-2,5 δισεκατομμύρια που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα και τι θα τους ταΐσουμε. Ε, χρειαζόμαστε ε, μία πολύ πιο πλατιά και ενδιαφέρουσα βάση διατροφική, ας πούμε. Δεν μπορούμε να τους ταΐζουμε όλους τσαμπάτας ε, και πρέπει να παράγουμε όλα αυτά τα τρόφιμα με πολύ πιο βιώσιμο τρόπο. Πολύ πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Σας ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι θα έχουμε τις ευκαιρίες όπως είπατε και σε άλλες περιπτώσεις να ειδωθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις ε, χαίρομαι που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και καλή τύχη στις προσπάθειές σας, ε, στις κοινέ μας προσπάθειες, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος.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 ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο εκθέσεις για 40 λεπτά. Δεν θα ξεπεράσουμε το χρονομιλία, ζητώ συγγνώμη. Η πρώτη έκθεση είναι το πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία. Ας την ξεπετάσουμε, ξεπετάξουμε. Αντί για τον κύριο Φλόρενς, μιλάει ο κύριος Λαβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Καρλ Χάινς Φλόρενς, δεν μπορεί να παραστεί. Ξέρουμε ότι η κυκλική οικονομία είναι περίπλοκο θέμα Μιλάει για... Υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα αξιών, είναι δυναμική. Χρειαζόμαστε μια πραγματική πεξίδα για να μα βοηθήσει εμά του πολιτικού, αλλά και τι επιχειρήσει, για να πάρουμε τι σωστέ αποφάσει για να ε, υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Το πλαίσιο παρακολούθηση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο γι' αυτό. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε επακριβώ ποια μέτρα επηρεάζουν και σε ποιο βαθμό. Ο στόχος του πλαισίου παρακολούθησης είναι να μας επιτρέψει να ελέγξουμε Εάν κατευθυνόμαστε σωστή κατεύθυνση ή αν πρέπει να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βασίζεται σε πλήρη στοιχεία και ολιστικούς δείκτες. Η Κομισιόν μας έδωσε αυτό που υποσχέθηκε. Μας έδωσε ένα πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία. Κατά την άποψή μου, με τους ε, δείκτες που έχουμε, έχουμε μια πρώτη απλώς απόπειρα για να φτιάξουμε τελικά την πηξίδα που πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να τους επικαιροποιήσουμε. Αυτή την άποψη το, τη συμμερίζονται και, και κάποια κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι η πρόταση θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε την πρόοδο ε, και την υλοποίηση όλων των στόχων και των δράσεων σε όλα τα σχέδια δράσεις ε, για την κυκλική οικονομία της Κομισιόν. Αλλά καλύπτει μόνο κάποια από τα σχέδια δράσης. Η βασική εστίαση είναι ε, στον κύκλο ζωής ε, και στην ανακύκλωση. Η φάση των αποβλήτων είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να αποκολουθείτε, αλλά και οι αρχικές φάσεις της αλυσίδα θα πρέπει να εκπροσωπείτε στο, στη δέσμη των δικτών. Το σχέδιο δράσης αφορά θέματα της αποτελεσματικότητας των πόρων και τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η, πρόληψη, η χρήση των δευτερογενών πρώτων υλών ε, ε, θα πρέπει να ενσωματώνεται ήδη στη φάση σχεδιασμού και παραγωγής Και δεν απεικονίζονται σωστά στη δέσμη των δικτών. Χρειαζόμαστε περισσότερους και καλύτερους δείκτες. Ένα άλλο θέμα είναι ε, η παραγωγικότητα των δικτών και των πρώτων υλών και οι δείκτες των πόρων συγγνώμη, και οι δείκτες ε, για την παραγωγικότητα των πόρων. Γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι δείκτες, ε, Κομισιόν, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Και επίσης, δεν υπάρχει η σύνδεση με το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης περίπου 12 του ΟΗΕ. Ε, βιώσιμη ε, παραγωγή. Ε, μπορούμε πολλά να πούμε ακόμα, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Θέλω η Κομισιόν να ξαναδεί την πρότασή της ή τουλάχιστον να την αναθεωρεί συχνά ε, και να αναθεωρεί και τους δείχτες για να είναι πιο κατάλληλοι. Αυτό, για αυτό να το κάνει, αυτό θα, πρέπει να συνεργαστεί πιο στενά με το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, γιατί έχουν πάρα πολλές εμπειρίες ε, και εφαρμόζοντας δείκτε κυκλικής οικονομία. Αυτά λέει ο κύριος Φλόρενς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τη διαβίβαση αυτού του μηνύματο από τον κύριο Φλόρενς. τώρα. Ο κύριος Λάινεν για λογαριασμό τη κυρία Μοναφέ. Ναι, το επόμενο μήνυμα που θα διαβάσω κι εγώ μέρος της συναδέλφου σε σχέση με αυτό το θέμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η εργασία αυτή τη Επιτροπή, δηλαδή για τη δημιουργία 10 δικτών σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, δεν ανταποκρίνεται πλήρω στην ανάγκη τη δημιουργία ενό σαφού και διαφανού ε, πλαισίου παρακολούθηση, το οποίο θα είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδο με σφαιρικό τρόπο. Ε, μάλιστα, υπογραμμίζουμε το πώς αυτοί οι δείκτες της ε, Επιτροπής θα πρέπει να εστιάζονται ειδικότερα στην ε, ε, δημιουργία των ε, απορριμμάτων και στην ανακύκλωσή τους. Ωστόσο, η προτεραιότητα εδώ θα πρέπει να είναι η πρόληψη της δημιουργίας αυτών των απορριμμάτων. Επίσης, η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει υπόψη της την ανάγκη του decoupling της αποσύνδεσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης αφενός και χρήσης πόρων και βιώσιμης κατανάλωσης αφετέρου. Οπότε, ρωτούμε την Επιτροπή ε, έχει ε, λάβει υπόψη της ε, τα αποτελέσματα της πλατφόρμας σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών και πώς σκοπεύει να τα συμπεριλάβει στο πλαίσιο παρακολούθησης. Επίσης, δεν υπάρχει ένας δείκτης το οποίο μας ελειπτεί σε ό,τι αφορά την παραγωγική χρήση των πρώτων υλών. Επίσης, δεν υπάρχει ένας δείκτης σε ό,τι αφορά τη δρομή της κυκλικής οικονομίας στην επίτευξη των στόχων της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, αλλά επίσης δεν υπάρχουν και οριζόντιοι δείκτες οι οποίοι θα μετρούν τις συνέργειες ανάμεσα στα μέτρα τη κυκλική οικονομίας και άλλες πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η βιοοικονομία και η πολιτική συνοχή. Εδώ δράτω με ευκαιρίε να θέσω ε, το συμπληρωματικό ερώτημα προς την Επιτροπή ως προς το γιατί δεν ε, δημιουργήσει ένα ξεχωριστό δίκτυο ο οποίος θα μετρά την ε, συγκεκριμένη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόιτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 12 σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση. Και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υπογραμμίζουμε την ανάγκη η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να θέσει να, εφαρμόσει δράσεις ε, για ε, ε, εφαρμογή συλλογικών μέτρων και θα θέλαμε να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των δικτών, των δικτών και προκειμένου να συμπληρωθούν με τους δίκτες που αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος, τον κύριο Λάνο και την κυρία Μποναφέ. Κύριος Ντεμεσμάχερ. Α, όχι, δεν είναι πάνω στην αίθουσα. Ποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Θα δώσω τότε το λόγο στην κυρία Λαντεφούτζη από την Επιτροπή για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα. Να πω καταρχήν ότι χαιρετίζουμε ε, το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας ε, για, την, ε, για το πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας και ε, συμμεριζόμαστε την άποψή σας ότι δηλαδή πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή σας για τα σχόλια που έκανε. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι συμφωνούμε και εμείς ότι η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και η παρακολούθηση των σχετικών τάσεων είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής ε, ε, τις προτεραιότητες που θα πρέπει να ιεραρχήσουν και τους τομείς τους οποίους θα χρειαστεί ενδεχομένω ε, περισσότερη δράση. Εμείς λοιπόν θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία ενός πολύ απλού αλλά και αποτελεσματικού πλαισίου. Ε, παρακολουθήσεις και προσπαθούμε εδώ να φτάσουμε σε μια ισορροπία ανάμεσα στο να καλύψουμε όσα μπορούμε αλλά και από την άλλη πλευρά ε, να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Και γι' αυτό η δική μας προσέγγιση ήταν επιλεκτική. Ε, προσπαθώντας όμως ταυτόχρονα να καλύψουμε τα τέσσερα θεματικά ε, πεδία του σχεδίου δράσης για την κλική οικονομία του 2015. Και εδώ έρχομαι Ε, σε ένα-δυο συγκεκριμένα ερωτήματα που μου έθεσαν τα αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Ε, τέθηκε λοιπόν επανειλημμένα το ερώτημα του γιατί η αποτελεσματική χρήση των πόρων δεν ελήφθη υπόψη του. Εμείς θεωρούμε πως η, παραγωγή, η, αποτελεσματική χρήση αλλά και η παραγωγικότητα σε σχέση με τους πόρους και τις πρώτες ύλες είναι σημαντικά, αλλά ακριβώς στο πλαίσιο της ισορροπίας που ανέφερα ε, πριν δώσαμε περισσότερη έμφαση σε ορισμένες πτυχές της κυκλικής ε, οικονομίας, δηλαδή ε, στην βιώσιμη κατανάλωση, στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και άλλους τομείς. Ωστόσο, Ε, δημιουργήσαμε δύο ε, διαφορετικά scoreboards, ε, δηλαδή πίνακες βαθμολόγησης αν θέλετε, με διαφορετικό στόχο και έτσι λοιπόν αυτές οι δύο δέσμες αν θέλετε δικτών έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα μία προς την άλλη και υπάρχουν μια κάποιες επικαλύψεις. Από την άλλη πλευρά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε το ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε την επιτεύξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Να πω εδώ ότι τέσσερις δείκτες από αυτούς που έχουμε εδώ είναι κοινή με αυτού που χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο τη δέσμη ε, των στόχων βιώσιμη ανάπτυξης για την επίτευξη συγκεκριμένα των ε, στόχων 11 και 12. Σε ό,τι αφορά τώρα, το ερώτημα που τέθηκε σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση του decoupling. Ναι, πράγματι υπάρχουν μια σειρά δικτών που σχετίζονται με τα απορρίμματα, με τα απόβλητα ε, και εδώ θα πρέπει βέβαια να εξετάσουμε πάντοτε το πού έχουμε την απαραίτητη ποιότητα ε, των δεδομένων. Ε, δηλαδή βλέπουμε το ΑΕΠ και την σχετική κατανάλωση αγαθών, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας και τον οικονομικό αντίκτυπο σε επίπεδο κλητής οικονομίας. Αυτά από την πλευρά μου και σας ε, ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω με ενδιαφέρον το τελικό ψήφισμα. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Κλείνουμε και με αυτό το σημείο τη σα διάταξη και περνάμε στο τελευταίο σημείο τη ε, ημερήσια διάταξη, η νόσο ΛΑΙΜ, δηλαδή η βορελίωση. Και εξετάζουμε εδώ ένα ε, σχέδιο ψηφίσματο. Να δώσω λοιπόν το λόγο ε, στου αισιόδου συζητητέ, με πρώτο τον κύριο Πέτρελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η αρρώστια που την έμαθα από πρώτο χέρι, από μένα. Έχω δηλαδή προσωπική εμπειρία από αυτή την αρρώστια. Είναι μια περίπλοκη αρρώστια. Γίνεται όλο το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται αυξάνεται, που νοσούν αυξάνεται και από ό,τι φαίνεται η κλιματική αλλαγή έχει συνεισφέρει στην ε, πλατιά εξάπλωση της αρρώστιας αυτής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγνωστεί αυτή η αρρώστια. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι οι ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί από αυτή την αρρώστια, από την νόσο του Λάιμ. Και πολλοί ε, ασθενείς ε, θεωρείται ότι νοσούν από κάτι άλλο χωρίς να γνωρίζουν ότι απλώς έχουν βορελίωση. Από ό,τι φαίνεται, αυτό δείχνει ποια είναι η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τη συνεργασία. Έχουμε κάποιες πρακτικές που είναι εξατομικευμένες όμως, μεμονωμένες, αλλά δεν έχουμε μια κοινή προσέγγιση για την αρρώστια αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δούμε τι τεχνογνωσία έχουμε ο καθένας μας, να υποφεληθούμε και να έχουμε πιο κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ για να προσεγγίσουμε καταρχά την αρρώστια. Ξέρουμε ότι η χρηματοδότηση, μια επιπλέον χρηματοδότηση είναι εκ των ονουκάνευ, ούτω ώστε να έχουμε μεθόδους ε, εντοπισμού και θεραπείας της ασθένεια. Ερευνητικά κονδύλια, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν, είναι πολύ σημαντικά. Είμαστε οχτώ συντάχτες εδώ ε, του κειμένου αυτού της προφορικής ερώτησης που έχουμε απευθύνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί κάνουμε αυτή την προφορική ερώτηση, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε μια μεγαλύτερη έμφαση σε μια κοινή προσέγγιση ε, και αυτό θα ήταν ε, πολύ πιο χρήσιμο για πολλούς ασθενείς μακροπρόθεσμα ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το χρωστάμε στους πολίτες μας αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος κυρία Σίπελ, τώρα ο κύριος Θανασέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σας πω και δύο λόγια από τη συνάδελφο τη Τατσιάνα Σάρμπου για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα, τη βορελίωση. Τα στατιστικά δείχνουν υπάρχουν ελάχιστα μικροπράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την πρόληψη αυτής της ασθένειας, αλλά αυτά τα μέτρα δυστυχώς δεν λαμβάνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν εκστρατείε πρόληψης, ιδίω σε περιοχές ε, που είναι πιο ε, εκτεθειμένες ε, σε τσιμπήματα από τσιμπούρια. Γι' αυτό ακριβώ και ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να προωθήσουν αυτέ τι ε, εκστρατείε και να παρέχουν και τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για να ε, γίνουν οι εκστρατείε. Επίση, να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία διάγνωση τη νόσου του Lyme και ε, τα τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται δεν είναι πάντα ακριβή. Χρειαζόμαστε βασικό συντονισμό και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και ε, ε, να υπάρχουν και συγκεκριμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Επίσης, πιστεύω ότι με το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για έρευνα στον τομέα αυτό, για εναλλακτικέ θεραπείες και πολύ πιο ακριβές ε, διαδικασίες δοκιμών. Ε, η μικροβιακή εντοχή είναι όλο ένα και πιο κοινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καλύτερος τρόπος ε, να θεραπευτεί η συγκεκριμένη νόσος είναι με αντιβιωτικά. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην σύνταξη του ψηφίσματος για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βυσνιεύσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Η βορελίωση είναι αυξανόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη και πρέπει να σας πω ότι στην Πολωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα ο αριθμός των περιπτώσεων αυξήθηκε ε, στο δεκαπλάσιο. Σε όλη την Ευρώπη μπορεί να έχουμε και ένα εκατομμύριο ασθενείς που έχουν νοσήσει από τη ε, βορελίωση. Νομίζω λοιπόν ότι πραγματικά σωστά λέμε ότι πρόκειται για μια σιωπηρή επιδημία. Και γιατί είναι σιωπηρή επιδημία, διότι αυτοί οι οποίοι πάσχουν από την νόσο ε, πολλές φορές ε, δεν λαμβάνουν ε, ακριβή διάγνωση έχουν κάποια συμπτώματα, αλλά δεν έχει ε, διαγνωστεί ως βορελίωση αυτό το οποίο έχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ελπίζω να υπάρχει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να βρούμε κονδύλια να υποστηρίξουμε έρευνα η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει και να έχουμε πιο αποτελεσματικές μεθόδους ε, θεραπείας ε, της νόσου ώστε να γίνεται και πιο έγκαιρη διάγνωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ πολύ τους με την προσέγγιση των συντακτών, διότι υπάρχει πραγματικά ανησυχία. Προσφάτως ε, έγινε μια συνεδρίαση για την επιδημιολογία στη Γαλλία και υπήρχαν πάρα πολλοί ε, διαδηλωτέ μπροστά από την αίθουσα, διότι για αυτούς ε, είναι έγκλημα το γεγονό ότι δεν αναγνωρίζεται η νόσο αυτή και είναι πραγματικά πρόβλημα η διαγνωσή της. Τι ζητούμε λοιπόν, ζητούμε εναρμόνιση των κριτηρίων. Πρέπει τα κριτήρια να είναι ίδια σε κάθε χώρα, διότι αλλιώ πώ θα αξιολογήσουμε τους πάσχοντες. Αναφερόμαστε ε, σε 650.000 με 850.000 στην Ευρώπη, αλλά ε, τα ποσά αυτά κυμαίνονται στον ΠΟΗ γιατί δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Και επίσης έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών ε, υπάρχει, ε, για παράδειγμα, στο τεστ Ίζα και το Western Blot ε, στη Γαλλία, ενώ σε άλλες χώρες γίνονται άλλα τεστ. Επομένως, πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση, να ξέρουμε ποια είναι τα καλύτερα τεστ διάγνωσης και κατόπιν η θεραπεία. Διότι η θεραπεία ε, για κάποιους είναι μια συγκεκριμένη, σε κάποιους προσφέρονται αντιβιωτικά, ε, κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολλά αντιβιωτικά γιατί μετά έχουμε μικροβιακή αντοχή ε, και η ψηλή ε, αρχή ε, υγείας ε, στην Γαλλία λέει ότι θα πρέπει να δοθούν τουλάχιστον αντιβιωτικά για 20 μέρες και μετά θα δούμε τα κλινικά συμπτώματα και τις συνέπειες. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ευρώπης είναι να συστήσει ομάδες εργασίας, να φροντίσει να υπάρξει ένα δίκτυο συνεργασίας για να μπορέσουμε να υπάρχει εναρμόνιση των κριτηρίων, να ξέρουμε ε, ποια είναι τα τεστ διάγνωσης και μάλιστα ποια ε, ε, αποζημιώνονται από τις ε, ασφαλιστικές εταιρείες γιατί κάποιοι πηγαίνουν και σε άλλες χώρες και κάνουν, διάγνωση, ε, κάνουν τεστ διάγνωσης και δεν αποζημιώνονται και επίσης με εντυπωσιάζει πως οι άνθρωποι δεν νιώθουν καλά, πιστεύουν ότι πάσχουν από Lyme, δεν πρόκειται τελικά για λάιμ, πρέπει κάπως να γίνεται μια σωστή διάγνωση. Η κυρία Ρίστο, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ Ε, όπως και οι υπόλοιποι, γνωρίζουμε δεκάδες ασθενείς. Οι οποίοι έχουν χάσει πραγματικά τον μπούσουλα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ε, είναι τεράστιο θέμα αυτό και συχνά το αφήνουμε τελευταίο στην ατζέντα μας, στο τέλος της συνεδρίασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ήμουν και εγώ όπως ε, με τη Μισελ στη Γαλλία ε, και στο Λουξεμβούργο για μια διάσκεψη ψηλού επίπεδου με ασθενείς, με γιατρούς και εμπειρογνώμονες ε, με πρωτοβουλία μιας βελγικής ε, οργάνωσης που λέγεται Time for Lime Υπάρχουν στην Ευρώπη και στο Βέλγιο διάφορες οργανώσεις που μας έχουν στο στόχαστρο, βλέπουν τι κάνουμε εδώ πέρα και βλέπετε ότι παρά τις δυσκολίες προχωράμε. Είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι. Η Λούση είναι εδώ παρούσα, η οποία ήθελε να συμμετάσχει στις ε, συνεδριάσεις μας, παρότι δυσκολεύεται να μετακινηθεί. Ε, μας ακούει λοιπόν και θα προσπαθήσει και εκείνη να μεταδώσει ας πούμε και να διαδώσει αυτά που κάνουμε εμείς. Ε, γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, βλέπουν τείχου να υψώνται απέναντί του. Δεν τους καταλαβαίνουν οι κλασικοί γιατροί, δεν καταλαβαίνουν, δεν, τους, ε, δεν βλέπουν ε, το πρόβλημά τους. Επίσης, τα τεστ για τον ιό ε, δεν είναι πολύ αξιόπιστα. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο ασθενεί στην Ευρώπη που έχουν την ασθένεια του Lyme. Συχνά του τσίμπησαν και δεν το κατάλαβαν εγκαίρω. Ε, συχνά αυτά τα τσιμπίσματα και η αρχή τη μόλυνση ε, δεν ε, πονάνε ούτε ενοχλούν καθόλου, ούτε καν σε τρώνε αυτά τα τσιμπίσματα. Ε, επανέρχομαι λοιπόν στο κείμενο το οποίο έχουμε μπροστά μα, το οποίο είναι φιλελεύθερο. Στην παράγραφο 11 ζητάει να πάμε πιο μακριά σε ό,τι αφορά την ανείχνευση, τον εντοπισμό τη ασθένεια. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη πολύ συγκεκριμένα, γιατί είναι δική του αρμοδιότητα, να γίνει μια κλινική εξέταση. Ωστότε η, δια, οι γιατροί να μπορούν να εντοπίζουν την ασθένεια του Lyme, ακόμα και σε περίπτωση που τα τεστ, τα σερολογικά είναι αρνητικά. Είναι πολύ σημαντικά. Τηλεγραφικά τα λέω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έτσι, να αναφέρω και άλλα δύο σημεία, πολύ σημαντικά του σχεδίου ψηφίσματο. Καταρχά, το θέμα τη έρευνα, σημείο 3 και 4. Η Κομισιόν παίζει σημαντικό ρόλο γιατί χρηματοδοτεί με 16 εκατομμύρια ευρώ την ε, έρευνα για πρόορη ανείχνευση ε, εντοπίζουμε κατευθείαν το βακτηρίδιο δηλαδή και να τεθεί στην αγορά ε, ένα πιο αξιόπιστο τεστ, ζητάμε να πάει ακόμα πιο μακριά στα πλαίσια του ένα, ένα του προγράμματος ε, έρευνας, περισσότερα κονδύλια επίση, πιο μακριά και καλύτερα σε ό,τι αφορά επίσης την συνεργασία, τη δικτύωση. Θα πρέπει, δεύτερο σημαντικό σημείο, η αρρώστια αυτή να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατόν στον Ευρωπαϊκό ε, Κατάλογο Μεταδόσιμων Ασθενειών, Μεταδοτικών Νοσημάτων, σημείο 14 και 15, Ευρωπαϊκό Δίκτυο, που θα επιτρέπει στους ασθενείς να υποφεληθούν ε, από σύστημα υγείας ε, καλό, διαρθρωμένο. Το ψήφισμά μας σε αυτό το επίπεδο είναι το πρώτο για την ασθένεια του Lyme. Καταγγέλει την, τον κομφορμισμό και συντηρητισμό πολλών ιατρικών συλλόγων κτλ. καταγγέλει εντό εισαγωγικών. Ε, γιατί εμείς ω Επιτροπή υγεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να είμαστε δίπλα στους ασθενείς και με την πλευρά των ασθενών. Ευχαριστώ, κυρία Αχής. Η κυρία Ντονανού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω συνεισηγήτρια, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να περιοριστεί στο να δημοσιεύει για αυτό το θέμα κατευθυντήριε γραμμές που θα βασίζονται στις καλύτερες πρακτικές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση των γενικών παθολόγων. Ο στόχος είναι να διευκολύνουμε την καλή διάγνωση και την ανείχνευση της ασθένειας του Lyme. Επίση, κατευθυντήριε γραμμέ θα μπορούσαν να δημοσιευθούν για να ενημερώνονται καλύτερα ε, για το βαθμό αξιοπιστία των σερολογικών τεστ και των μη συμβατικών ε, θεραπείων. Ε, επίσης υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης ό,τι αφορά την αξιολόγηση ε, του μεγέθου ε, του ιατρικού λάθους ε, που πέφτουν θέματα διάφοροι ασθενείς και κυρίως συχνά βλέπουμε ανθρώπους που μετακινούνται από τη μια χώρα στην άλλη, περνάνε τα σύνορα για να λάβουν θεραπεία για την αρρώστια του ΛΑΙΜ. Ο ρόλο τη Κομισιόν θα μπορούσε να περιοριστεί στο να συλλέγει τι περισσότερε δυνατέ πληροφορίε για τι μεθόδου ανείχνευση ή για τι θεραπείε που χορηγούνται στα κράτη-μέλη χωρίς όμως να σφετερίζεται το ρόλο των κρατών μελών. Η Κομισιόν θα μπορούσε να ενθαρρύνει δηλαδή εκστρατείε ευαισθητοποίηση των πολιτών ε, στους κινδύνους ε, της ασθένεια αυτής μετά από τσιμπήματα του κρότονα και ε, να μην ξεχνάμε ότι η, η ασθένεια εμφανίζεται πολύ μετά ε, και με πολύ διαφορετικά συμπτώματα κάθε φορά από το τσίμπημα. Επίση, ε, με διαφάνεια θα πρέπει ε, η Κομισιόν να λέει στα κρατη τα επιστημονικά συμπεράσματα, γιατί έχουν επενδυθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα τη ασθένεια του Λάιν και να εκπονηθεί ένα και να ενημερώνει για τον εμβόλιο που υπάρχει. Πρέπει να δούμε, χρησιμοποιήθηκαν καλά αυτά τα χρήματα, έχουμε δικαίωμα σε κάτι τέτοιο. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα ήθελα να εισαγάγω μέσω των τροπολογιών μου. Ευχαριστώ. Κυρία Γκοντίν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι που επιτέλους μιλάτε για αυτό το θέμα. Η ασθένεια του Λάιμ επί χρόνια ήταν ο φτωχός ασθενής ε, των, ε, ε, στην επιδημιολογία. Ε, επιτέλους τώρα κάνουμε μια κοινή σκέψη, ένα κοινό προβληματισμό για να συντρέξουμε τους ε, πάσχοντες. Ξέρουμε ότι η εξάπλωση των ε, τσιμπουριών και των τσιμπημάτων είναι άμεσα υπεύθυνη για την εξάπλωση της ασθένειας αυτής στην Ευρώπη. Εντάξει, γιατί μιλάμε κυρίως για ένα εκατομμύριο περιπτώσεις κρούσματα. Επιπλέον έχουμε την αδράνεια έλλειψη μέσων και αδιαφορία από τις δημόσιες αρχές για αυτή την αρρώστια της υπαίθρου. Και αυτό όμως παρά αυτά δεν εξηγείται από το γεγονός ότι έχουμε τόσα πολλά τσιμπήματα και εξάπλωση της ασθένειας. Για να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες θα πρέπει να δούμε ε, το γιατί πεθαίνουν μαζικά ε, τα πτηνά στην Ευρώπη, τα πουλιά στην Ευρώπη που τρώνε τσιμπούρια. Ε, η γενική χρήση ε, ζυζανιοκτώνων και φυτοφαρμάκων ε, οδήγησε σε μείωση των ε, θρεπτικών πόρων για τα, για τα πουλιά και μια αντίδραση, μια αντίσταση μάλλον των τσιμπουριών ε, λόγω αυτών των χημικών. Ε, τα προβλήματα υπάρχουν κυρίως στις περιοχές Υπέθρου και δίπλα στην Υπέθρου. Ε, επίσης, Εκεί δεν έχουμε και αρκετά καλού ή αρκετά ενημερωμένου γιατρού στι περιοχέ αυτέ ε, υπαίθρου. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα ε, ανείχνευση ε, και πρόσβαση ε, ε, στην περίθαλψη. Αυτά είναι προτεραιότητα θέματα. Έχω την αίσθηση ότι με αυτή την αρρώστια δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Οι γεωργοί, οι γεωργοί δυσκολεύονται να αναγνωριστεί αυτή η αρρώστια ω επαγγελματική ασθένεια. Οι ασθενεί συχνά αντιμετωπίζουν το ιατρικό λάθος, γιατί δεν υπάρχουν ούτε ειδικοί γιατροί, ούτε πληροφορίες αρκετές, δεν υπάρχουν αρκετά μέσα για να βρεθεί κατάλληλο, ε, κατάλληλη θεραπεία και φάρμακο για αυτή την ασθένεια. Για, αυτή, ακριβώς την, ε, για αυτούς τους λόγους προσυπογράφω αυτή την ε, προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν, περιμένω απαντήσεις για να τις διαβιβάσω στους πάρα πολλούς ασθενείς της εκλογική μου περιφέρειας. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόλνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Για να απαντήσετε στα ερωτήματα ή να, να σχολιάσετε τις ιδέες που ακούστηκαν. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε από την Επιτροπή σας, ε, για το σημαντικό αυτό το ζήτημα και για τα σχόλια που έδιναν αλλά και τα ερωτήματα που τέθηκαν. Πράγματι, ε, νόσος του Λάιμ είναι μία από τις σημαντικότερες μεταδοτικές ασθένειες στην Ευρώπη και ε, η πιο σημαντική ασθένεια που μεταδίδεται από τσιμπούρια. Και η επιδημιολογία εδώ είναι ασαφής ε, γιατί ακριβώς υπάρχει αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την ε, διάγνωση και τα συμπτώματα που παρουσιάζει αυτή η ασθένεια αλλά και λόγω της διαφοράς των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της νόσου Μέχρι στιγμή αυτή η ασθένεια δεν ήταν υποχρεωτικό να αναφέρεται ε, και οι αναφορέ δηλαδή των δεδομένων γινόντων ήταν μόνο από ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ενημερώσω σε σχετικά με μια νέα εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά σοβαρέ απειλέ για την υγεία που θα υιοθετηθεί αύριο. Εκεί λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των μεταδοτικών νόσων, θα συμπεριλάβουμε και τις ασθένειες που θα πρέπει να καλύπτονται από την ε, επιδημιολογική παρακολούθηση με βασικούς ε, δείκτες και θα περιλάβουμε ασθένειες οι οποίες έχουν ε, προκύψει πρόσφατα, όπως για παράδειγμα και η προλίωση, δηλαδή η νόσος του ΛΑΕΜ. Οι σχετικές λοιπόν πληροφορίες και τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης για το οποίο είναι αρμόδιο και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την πρόληψη των Ασθενειών οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα ε, διαβιβάζουν λοιπόν στο μέλλον αυτές τις πληροφορίες στο κέντρο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο, συγκεκριμένο, ε, συμφωνισμένο ορισμό πράγμα το οποίο θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης αυτής της ασθένειας. Ε, και βέβαια αυτή η απόφαση ε, λήφθη με βάση τα νέα δεδομένα που, ε, των οποίων έλαβε γνώμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω ήδη αναφέρθηκε, και με βάση τα νέα δεδομένα που έχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Ασθενειών. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλε δράσει, όπω δηλαδή περισσότερη επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του ευρέω κοινού, το κέντρο εργάζεται και επί αυτών των ζητημάτων και ετοιμάζει μια δημοσίευση σε ό,τι αφορά τη νοστουλά με την προλίωση και έχει δημοσιεύσει ε, και ένα ε, kit ενημερωτικό σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, φυλάδια, παρουσιάσεις, πόστερ, αφήσει. και κάνει και κάποιες εργασίες σε ό,τι αφορά τις διαγνωστικές μεθόδους και αναθεωρεί και τις διαθέσιμες πληροφορίες για αυτό το ζήτημα, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο του ψηφίσματος σας. Και, αναφέρθηκε και η περιοχή Ρίτς αλλά και μία σειρά από άλλα project τα οποία είναι σημαντικά για την ε, ε, νόσο του ΛΕΜ. Ε, και αυτό εντάσσεται στις προσπάθειες που γίνονται για καλύτερη, ε, για καλύτερη ε, διάγνωση αλλά και ανάπτυξη εμβολίου για το ΛΑΕΜ μέσω και προώθηση του σχετικού προγράμματος πλαισίου 7 και της σχετικής χρηματοδότησης αλλά και στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Μία σειρά από αυτά τα project ήδη έχουν αναφερθεί. Αυτά από την πλευρά μου και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω περαιτέρω ερωτήματα σε σχέση με αυτές τις δράσεις της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτησή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 26 Ιουνίου 11 η ώρα και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό ολοκληρώνεται η συνεδρίαση για σήμερα. Καλή σας όρεξη.